Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα θα πρέπει να συνηθίσετε σε άλλη φωνή. Λυπούμε, αλλά ο Αλένα Μασούρ έχει μπλοκαριστεί σε μια διαδήλωση. Δεν είναι ότι συμμετέχει στη διαδήλωση, και δεν ξέρω καν το περιεχόμενο της διαδήλωσης, πάντως μου είπαν ότι έχει μπλέξει σε μια διαδήλωση, έχει κολλήσει το αυτοκίνητό του και προς το παρόν κολλείεται να φτάσει γέρο στην Επιτροπή μας, γι' αυτό θα ξεκινήσω εγώ. Όπως είχαμε προβλέψει θα αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Ας περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμό 4 της Συντόνια Γεντζογεύσκα. Δεν θέλει το λόγο η συγγήτρια, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Έχουμε μια τροπολογία. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές ψηφίζουμε τώρα την έλλειψη διόρθωσης ποιος είναι υπέρ, κατά Φαίνεται ότι έχουμε λιγότερες αρνητικές ψήφους εδώ. Αποχές. Καλά, εγκρίνεται. Είμαστε υπέρ, υπέρ. Λυπάμαι, ε, έγινε ένα λάθος συντόνια. Επόμενο σημείο. Έκθεση Μπάρμπαρα Ματέρα. είπαν ότι προηγείται στην ψηφοφορία έκθεση Καρλ Χάγκλουντ. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες για την έκθεση Χάγκλουντ. Τροπολογία 1 ε, έχει αποσυρθεί. Απο, ε, τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Warren. Κατά. Αποχές. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ. Τροπολογία 8 με 23. 8 23. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε ομαδών. Υπάρχει αντίρρηση να ψηφιστούν από κοινού. Όχι. Οπότε τις ψηφίζουμε μαζί. πολλά λάθη κάνουμε σήμερα. Οχτώ με 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Επόμενο θέμα. Τροπολογία 2 για την επιλογή σκέψη 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Η υπόλοιπη υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ του εισηγητού είναι η τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 στην ιδεολογική σκέψη 16. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον διορθώνει πρόεδρος. Τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 27-28 πανομοιότυπες, ποιος είναι υπέρ. Κατά. <coughs> Αποχές. Μία αποχή. Η υπόλοιπη κατά. Τροπολογία 5. Στην αιτιολογική σκέψη 18. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μία αποχή Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ομόφωνα. 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφος κατά. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μία αποχή <clears throat> εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μια αποχή αλλά απορρίπτεται. Ε, ομόφωνα, ομόφωνα, ομόφωνα. 35 <clears throat> υπέρ κατά απόχέ. με μια αποχή οι υπόλοιποι εγκρίνουν, 36 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ομόφωνα τελική ψηφοφορία ψήφι υπέρ της τροποποιημένης ε, εκθέσεως κατά αποχές με μία αποχή οι υπόλοιποι εγκρίνουν και συγχαρητήρια Ματέρα. Also sofort, sofort. Es gibt. Η πρόεδρος, αμέσως. Δύο πράγματα μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα, δύο περιπτώσεις ας πούμε. Η τρίτη δεν τίθεται σε ψηφοφορία ακόμη, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε ακόμη όπως μόλις με πληροφόρησαν. Θα ακούσουμε όμως πρώτα την εισηγήτρια. Θα είμαι σύντομη κυρία Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση προπολογισμών σας είχα παρουσιάσει αναλυτικά το θέμα των τριών περιπτώσεων που θα συζητήσουμε τώρα, της Δανίας, τη ε, Γερμανίας και της Πορτογαλίας, που δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την υπόθεση Ρενό, όπου ζητείται κινητοποίηση του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, που είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί στο Ταμείο αυτό, διότι πρόκειται για βοήθεια ε, σε πάνω από 3.000 εργαζομένους και έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επομένως, η Επιτροπή Προεπολογισμών ε, μαζί με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, του Κοινοβουλίου ζητά διευκρινήσεις στους επικεφαλείς της Ρενό. Μέχρι να λάβουμε τις διευκρινήσεις αυτές, συμφωνούμε όλοι για την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι είναι πολύ σημαντικές και οι ψηφοφορίες που θα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη στο Στρασβούργο στη διάρκεια της Συνόδου για το μέλλον του του συγκεκριμένου ταμείου. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, φανεί από την ψηφοφορία ότι είμαστε ομόφωνοι και να προσπαθήσουμε να ε, διασκεδάσουμε όλες αυτές τις μικρές δυσκολίες και τους προβληματισμούς που προκύψαν από την οθότηση του ψηφίσματος του Πρόεδρου Μπερές. Θα θέλαμε να υπάρχει μια καλή πλειοψηφία στην Ολομέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν να ψηφίσουμε τρία, τρεις ε, περιπτώσεις την δανική, γερμανική και πορτογαλική θα αρχίσουμε με τη δανική υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες τις οποίες θα διεξέλθουμε τώρα η πρώτη υπαριθμών δύο ψήφι υπέρ παρακαλώ κατά παρακαλώ και αποχές εσείς είστε υπέρ μάλιστα έξι ψήφοι κατά εγκρίνεται κατά τα άλλα τροπολογία τρία υπέρ κατά με έξι ψήφους κατά εγκρίνεται από τους υπολείπους τέσσερα τροπολογία τέσσερα υπέρ κατά με επτά ψήφους κατά εγκρίνεται ωστόσο Α, ναι, ξέχασα να ρωτήσω ποιος απέχει της ψηφοφορίας. Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Όλοι νομίζω. Αποχές. Όλοι κατά. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Είναι σαφής η πλειοψηφία κατά. Αποχές, μια αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Υπαριθμόν 7 υπέρ. Κατά. Όλοι. Όλοι κατά. Αποχές. Καλά λοιπόν. Όλοι κατά. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές με μια αποχή. πέντε ψήφοι υπέρ, οι υπόλοιποι κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το τροποποιημένο κείμενο, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές, δύο αποχές, δύο ψήφι κατά, δύο αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Αλλά θα σας πω συγχαρητήρια, Μπάρμπαρα, όταν θα έχουμε τελειώσει και τα τρία. Η δεύτερη υπόθεση, η γερμανική υπόθεση τώρα. Δύο τροπολογίες, υπαριθμών δύο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μια αποχή, έξι ψήφοι υπέρ, υπόλοιποι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, έξι υπέρ. Υπόλοιποι κατά απορρίπτεται. Τελευταία ψηφοφορία, τελική μάλλον ψηφοφορία, υπέρ του συνόλου της εκθέσεως. Κατά. αποχές τρεις ψήφοι κατά δύο αποχές οι υπόλοιποι τάσσονται υπέρ εγκρίνεται λοιπόν τώρα η πορτογαλική περίπτωση όπου δεν υπάρχουν τροπολογίες ψήφοι υπέρ να το εγκρίνουμε δηλαδή όπως το προτείνει η κυρία Ματέρα κατά αποχές Τέσσερι αποχές, μία ψήφος κατά. Οι υπόλοιποι εγκρίνουν, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν Μπάρβαρα, και για τις τρεις περιπτώσεις που εγκρίθηκαν. Και ακολουθεί. Ακολουθούν μάλλον <clears throat> οι μεταφορές πιστώσεων. Okay. So we wait, and we, we hope that the Commission will wait to mm say. The Commission should wait for Okay. Also den ähm, Transfer Nummer 22, den werden... Το 22 δεν θα το ψηφίσουμε τώρα, διότι έχει σχέση με την περίπτωση Ρενό, που εκκρεμεί ακόμη. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα προχωρήσουμε στην 25 μεταφορά 25, η Σιδονία είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται λοιπόν. Υπαριθμόν 26 μεταφορά πιστώσεως. Η Σιδονία είναι υπέρ. Εκ των υπολείπων ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ουδής απέχει. Ωραία. Μία ψήφος κατά εγκρίνεται λοιπόν. Η υπαριθμόν 27. Είναι και η τελευταία ψηφοφορία που θα διεξαγάγω εγώ. Η Σιδωνία είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά μία ψήφο κατά, αποχές, κανείς. Καλά λοιπόν, εγκρίνεται και αυτή. Παραδίδω τώρα τα ενία της συζητήσεως στον πρόεδρό μας που μόλις κατέφτασε. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη και από τη Γιώτα και τους λοιπούς αλλά διεξάγονται διαδηλώσεις στους δρόμους των Βρυξελών και τελικά καθυστέρησα στην έλευσή μου από το σταθμό του τρένου. βασμένου λοιπόν τώρα ορισμένες μεταφορές πιστώσεων ακόμη και πρώτα η παριθμόν 23. Η Σιδανία είναι υπέρ. Κατά. Ε, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. Μεταφορά υπαριθμών 30. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Μία ψήφος κατά αποχές. Χωρίς αποχές εγκρίνεται. 32. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Για τις Κατά. Αποχές. Το ίδιο εγκρίνεται. 33. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Καλώς κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή η μεταφορά. Έχουμε και άλλες ε, ψηφοφορίες για μεταφορές πιστώσεων από προπολογισμό για τα λοιπά τμήματα, αλλά λίγο αργότερα θα σας πρότεινα να ψηφίσουμε τα σημεία αυτά, γιατί όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μία επιτροπή συνδιαλλαγής. Συνεδρίαση επιτροπή συνδιαλλαγής για το σχέδιο προπολογισμού του επόμενου έτους και μια και η κυρία Τρυπελίνη συγγήτρια συμμετέχει σε αυτή την συζήτηση προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις υπόλοιπες μεταφορές, περιμένοντας την εισηγητριά μας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι το σημείο 7, μια και παρίσταται ο Ράιμερ Μπέγκερ μπορούμε να το εξετάσουμε. Το σημείο 7 αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πολι... δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Δυστυχώς ο Ζαν Λιουκ Ντεάν μου ανακοίνωσε ότι θα απουσιάσει σήμερα. Κύριε Μπέγκερ, έχετε κάποια στοιχεία να μας μεταφέρετε. Σας υπενθυμίζω ότι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της νέας διαδικασίας που ε, συμφώνησε και εφαρμόζει η Πολωνική Προεδρία προβλέπει ανταλλαγή απόψεων πριν το πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που εγγενίασε τη συζήτηση αυτή και που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου. Ε, στις 12 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Στο τρίο των αντιπροσωπιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνταν από μια προσωρινή επιτροπή που απαρτίζονταν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, την πρόεδρο της Επιτροπής ΣΟΥΡ και τον βασικό μας ηγητή, τον κύριο Μπέγκε. Έκτοτε η ίδια ανακοίνωσε ότι θα οριστικοποιήσει την ε, σύνθεση της αντιπροσωπείας, αλλά από ό,τι ξέρω ακόμη δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, παρόλο που υποσχέθηκε το Προεδρείο ότι θα την, η συνδιάσκεψη των Προέδρων θα την ε, λάβει το συντομότερο δυνατό. Ως προς το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες συνεδριάσεις με το τρίο που θα εκπροσωπεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Τον Οκτώβριο δεν θα γίνουν συναντήσεις γιατί τον Οκτώβριο το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία της ε, διάσκεψης κορυφής. Ε, στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και οι δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων θα επικεντρωθούν και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τον Νοέμβριο να έχουμε και μια συνεδρίαση για μια γενική επισκόπηση των δύο πιο σημαντικών από δημοσιονομική άποψη πολιτικών, που είναι η πολιτική συνοχή και η κοινή γεωρική πολιτική. Και το Δεκέμβριο θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για το νέο σύστημα ιδίων πόρων. Στις 20 και 21 Οκτωβρίου, πέραν των διαπραγματεύσεων, αλλά για μεγαλύτερη διαβίστηση της συζήτησης, θα έχουμε και μια ε, πανευρωπαϊκή δημοσιονομική διάσκεψη. Το είχε ζητήσει και ο κύριος Γκαρίγκα και ήταν και το ψήφισμα που υιοθετήσαμε στην, στην Ολομέλεια μετά από πρώτη επιτροπή ΣΟΥΡ. Θα γίνει μια διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη με συμμετοχή των κυβερνήσεων, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσει υψηλού επίπεδου μεταξύ του Κοινοβουλίου, τη Πολωνική Προεδρία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν λάβω πιο λεπτομεριακές πληροφορίες θα τις ανακοινώσω. Από ό,τι ξέρω αναμένονται 80 περίπου εθνικοί βουλευτές γιατί έχουμε 40 κοινοβουλευτικά σώματα στις 27 χώρες μέλη, γιατί έχουμε πολύ συχνά δύο βουλές, ανά και κάτω βουλή, βουλή και γερουσία. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητήσει να εκπροσωπηθεί και από 40 ευρωβουλευτές. Ε, βέβαια αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, δεν εμπίπτουν σε αρμοδιότητές μου. Μόλις ενημερωθώ θα σας ανακοινώσω τις πληροφορίες και θα σας ενημερώσω και για τη συνέχεια φυσικά. Υπενθυμίζω λοιπόν το γενικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Ε, δεν ξέρω αν ο Ράιμερ έχει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, Ράιμερ. Θα είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου έχουν λάβει ένα σημείωμα από τη Γραμματεία σχετικά με τα ζητήματα που τίθεται υπό συζήτηση 12, που τέθηκαν μάλλον στις 12 Σεπτεμβρίου σχετικά με τη διάρκεια της δομή του προϋπολογισμού καθώς και το εργαλείο ευκαμψίας να επισημάνω ότι Ελπίζουμε βέβαια οι, επόμενοι, επόμενες προεδρίες, Δανική και Κυπριακή, θα συνεχίσουν την πορεία της Πολωνικής, με τη συνεργασία δηλαδή με το Κοινοβούλιο, ότι θα συνεχιστεί εντατικά αυτή η συνεργασία. Όσο πιο εντατικές γίνονται οι διαβουλεύσεις, τόσο μεγαλύτερη σημασία λαμβάνουν οι ε, συνεδριάσεις αυτές, προ δηλαδή του ε, Συμβουλίου, των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Φάνηκε πόσο σημαντικό είναι με την εντολή της Επιτροπής Σούρε που επιβεβαιώθηκε και από την Ολομέλεια να υπάρχει ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ισχύσει και για τις μελλοντικέ συζητήσεις με τις προεδρίες του Συμβουλίου καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από την διάσκεψη αυτή όπου η πρόθεση είναι Δανική και Κυπριακή Προεδρία να θέσουν παρόμοια θέματα επιτάπητος. Τον Νοέμβριο λοιπόν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα μιλήσουμε για διαρθρωτική και γεωργική πολιτική και το Δεκέμβριο για τους ιδίους πόρους αρχίζει λοιπόν το όλο να παίρνει κάποια κίνηση, να αρχίζει να κινείται. Το ερώτημα είναι πότε θα αρχίσουν οι πραγματικές διαπραγματεύσεις, δηλαδή πόσο προοδεύουν οι συζητήσεις και από την πλευρά του Συμβουλίου έτσι ώστε να μπορέσει να υποβάλει μια λογική ε, πρόταση στο Κοινοβούλιο. Αυτό θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους μη ε, δημοσιονομικές. Αν δηλαδή θα μπορέσουμε με λίγα λόγια μέσα από την κρίση αυτή να δώσουμε μια νέα όθηση στην ε, ευρωπαϊκή ενοποίηση με συμμετοχή και των Εθνικών Κοινοβουλίων όπου βέβαια οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή έχουν χαρακτήρα αντιπαραθέσεως Θα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει η Πολωνική Προεδρία στη συνεργασία μαζί μας να συζητήσουμε και μεταξύ μας εδώ με την ησυχία μας πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα προετοιμαστούμε για τις επόμενες διατοχικές συνεδριάσεις και ποια στρατηγική θα διαμορφώσουμε για τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο. Από τη σκοπιά του, της Επιτροπής Προϋπολογισμών ένα θέμα θα είναι σημαντικό. Πώς θα μπορέσουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο να συζητήσουμε το ζήτημα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να το συνδέσουμε με τα μεγάλα νομοθετικά πακέτα τα οποία θα ακολουθήσουν ώστε να βελτιωθεί και η ποιότητα του νομοθετικού έργου και στα διαρθρωτικά και αλλού γιατί όσο πιο δύσκολα γίνονται τα νούμερα τόσο πιο σημαντική γίνεται ως προϋπόθεση συνεκβανών η ε, ευκαμψία, η ευελιξία. Αυτά και να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ε, κατησχίσει και μέσα στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Ευχαριστώ Ράιμερ. Από όλες τις συναντήσεις που είχαμε τις τελευταίες μέρες με την Πολωνική Προεδρία, είτε με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, είτε με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Μπιεβίτς, ή με τον κύριο Γιάννη Δομινίκ, τον Υφυπουργό για τα θέματα προϋπολογισμού, το συμπέρασμά μας είναι ότι η Πολωνική Προεδρία δεν βιάζεται να περάσει στις ε, διαπραγματεύσεις, στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γιατί ε, βρίσκονται και μέσω προεκλογικής εκστρατείας στην Πολωνία. Οπότε περιμένουν να, να ολοκληρώσουν το γύρο τραπέζι και την ανταλλαγή απόψεων, αλλά μάλλον θα αφήσουν στην ε, Δανική Προεδρία τα εγγένεια των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ακόμη και στο Συμβούλιο, μεταξύ των Υπουργών, αλλά και με το Κοινοβούλιο. Οπότε υπάρχει και ένας άλλος άγνωστος χ. Στη Δανία την περασμένη εβδομάδα είχαμε τις βουλευτικές εκλογές και αναμένεται ο σχηματισμός ε, νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Οπότε και η Δανία θα διαμορφώσει τη δική της διαπραγματευτική θέση εν ώψη των επικείμενων διαπραγματεύσεων και φυσικά θα αναλάβει τις ευθύνες προεδρίας στο επόμενο εξάμεινο. Συνεχίζουμε τις επαφές με την δανεική μόνιμη αντιπροσωπεία εδώ και αρκετές εβδομάδες ε, ώστε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον μια συνεχή ροή πληροφοριών από τη δανεική κυβέρνηση. Πάντως, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μάλλον με αργούς ρυθμούς και κατά πάσα πιθανότητα σε αρχές του επόμενου έτους όχι πριν τι αρχέ του επόμενου έτου. Πάντως, όπως είπε και ο Ράιμερ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει υποβάλει τις νομοθετικέ βάσεις για τις πολιτικές που θα χρηματοδοτηθούν από την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 για την γεωργική πολιτική, την πολιτική συνοχή και τι άλλε σημαντικέ από δημοσιονομική άποψη πολιτικέ. Ώστε να έχουμε μια γενική εντύπωση και για τους νέους προσανατολισμούς των πολιτικών που φυσικά θα ακολουθήσουν την ε, κανονική νομοθετική διαδικασία αλλά και να γνωρίζουμε και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ε, βλέπω ότι ο, συντονιστής ε, το ΕΛΚ έχει χάσει τη θέση του. Είχαμε ένα μικρό επεισόδιο στην ε, συνεδρίασή μα. Είναι αρκετά δυσάρεστο αυτό το φαινόμενο. Χάνει κανεί την έδρα του. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ξαναβρήκε. Ή, αν... Ευχαριστώ το Ράιμερ για τις πληροφορίες. Ε, ε, επειδή είμαι από την αντιπολίτευση στη Δανία, μπορώ να σας πω ότι η νέα αντιπολίτευση Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ αρκετών κομμάτων για το πώς θα πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, οπότε θα δείτε ότι υπάρχει συνέχεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βεβαίως, η επόμενη χρονιά θα επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες και έχει δίκιο. Πλέον μένει να δούμε τι δομή, τι διαρθρωτικά ταμεία θα έχουμε στο μέλλον πριν αποφασίσουμε για το πλαίσιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει λογική στις διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι στο τέλος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν με τον κύριο Φανρόμπα και ίσως θα πρέπει να προετοιμαστούμε κι εμείς για να δούμε πώς θα είμαστε κι εμείς τμήμα των διαπραγματεύσεων στο τέλος. Βεβαίω αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πολύ καλή προετοιμασία για να έχουμε μια καλή εικόνα του τι ποσά θα έχουμε για κάθε πολιτική, ώστε να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλέ εκκρεμότητε ε, όταν θα φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θα καθίσουμε στο τραπέζι με τα κράτη-μέλη και όλοι θα ζητάνε επιστροφή χρημάτων. Θα έχει κάποιο ενδιαφέρον και αυτό. Ε, ευχαριστώ. Αν Εξάλλου, αν κατενόησα καλά, ο μελλοντικός, μελλοντικός πρωθυπουργός θα είναι η κυρία Τόρνινγκ Σμιτ στη Δανία. Άρα, παλαιά συνάδελφός μας, μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και σημαντικό μέλος της συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης. Μπορεί κανείς λοιπόν να υποθέσει ότι η γενική κατεύθυνση που θα δώσει θα είναι μάλλον ευνοϊκή υπέρ του ευρωπαϊκού πνεύματος. Φυσικά αυτό είναι καθαρά δανέζικη υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάντως και προτείνω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό που έτσι και ήταν μόνο για ενημέρωση. Στο μεταξύ έχει έλθει η κυρία Τρίπελ, Έλγα Τρίπελ, που ήταν απασχολημένη αλλού στη συνδιαλλαγή. Ας, εάν είστε έτοιμοι, Χέλγα, ας ε, ψηφίσουμε τις μεταφορές πιστώσεων. Έχετε ορισμένες που μας προτείνετε. Ψηφίσαμε ήδη τις ε, ε μεταφορές πιστώσεων της ε, Σιδονία και νομίζω ότι έχουμε ακόμα τρία σχέδια μεταφοράς πιστώσεων για άλλα θεσμικά όργανα εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν τα πρώτα. Οι λοιποί συντονιστές και μέλη της ε, αντιπροσωπείας μας έχουν, έχουν έλθει και μόλις είστε έτοιμοι, αν θέλετε, να τις ε, θέσουμε σε ψηφοφορία. Η Επιτροπή Περιφερειών. Έχουμε την μία μεταφορά πιστοσύνη για την Επιτροπή Περιφερειών και η δεύτερη για το ελεγκτικό συνέδριο. Χέλγα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την πρώτη μεταφορά. Η πρώτη μεταφορά είναι μεταφορά πληροφοριών που ζητήσαμε από την Επιτροπή Περιφερειών. Γιατί οι διαδικασίες πρόσληψης στην Επιτροπή Περιφερειών δημιούργησαν τεράστιο κόστος ό,τι αφορά ε, τα ταξιδιωτικά έξοδα, τα επιδόματα κτλ. Οπότε θέλουμε μεταφορά πιστώσεων 24.000 ε, ευρώ από τη δημοσιονομική ε, γραμμή για την ανταλλαγή ε, υπαλλήλων, ε, δόματα υποτροφίες από τα διάφορα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Εγώ δεν έχω αντίρρηση ως προς τη ε, μεταφορά πιστώσεων που έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Περιφερειών. Καλώς. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς που βρίσκει σύμφωνη την εισηγητριά μας. Κατά. Μία ψήφος κατά αποχές, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη μεταφορά πιστώσεων για το ελεκτικό συνέδριο. Η κυρία Τρίπελ. Θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ δύο μεταφορές πιστώσεων ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνεδρίο ζήτησε μεταφορά 60.000 ευρώ από τη δημοσιονομική γραμμή αμοιβών των, ε, δημοσίων, των ε, μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων από την γραμμή για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Γιατί το ελεκτικό συνέδριο χρειάζεται περισσότερους μεταφραστές εξωτερικούς, γιατί οι εσωτερικοί μεταφραστές έχουν ανακυκλωθεί θα γίνουν ε, μέλη του ελεκτικού συνεδρίου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν, είναι δικό μας θέμα. Το δεύτερο αφορά ενίσχυση του, της δημοσιονομικής γραμμής για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για 20.000 ευρώ. Οι πιστώσει αυτές θα αφαιρεθούν από τη δημοσιονομική γραμμή του Ελεκτικού Συνεδρίου για την παραγωγή και έκδοση της επίσημης εφημερίδας και θα πρότεινα και πάλι να δεχθούμε τις δύο μεταφορές πιστώσεων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε από κοινού. Ωραία. Ποιος είναι υπέρ των δύο μεταφορών πιστώσεων για το ελεκτικό συνέδριο. Κατά. Μία ψήφο κατά. Αποχές εγκρίνονται οι δύο μεταφορές πιστώσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Καλώς, ολοκληρώσαμε τις μεταφορές πιστώσεων και τις ψηφοφορίες. Έλγα, παρακαλώ. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το σημείο 6 της της διάταξης. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμό 5 για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έλγα, θα μπορούσατε λοιπόν να μα παρουσιάσετε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού παριθμό 5, γιατί ξέρω ότι είχατε πολλέ επαφέ. Πείτε μα παρακαλώ. Τι εντύπωση αποκομίσατε, η κυρία Τρίπελ. Έχω ήδη διευκρινίσει τις θέσεις μας ε, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση προπολογισμού για τον Ευρωπαίο Επόπτη θεωρώ ότι αυτό είναι ίσονο σημασία και δεν θα έπρεπε να αναφέρεται σε σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Επιπλέον, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κατεπίγους ανάγκη να ε, ε, περάσουμε στην τροποποίηση του σχεδίου DESP ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το 2011 από τώρα. Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει στον επόμενο προϋπολογισμό και να μην γίνει τώρα με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Αν επιμένετε θα μπορούσα να σας δώσω και κάποιες επιπλέον πληροφορίες επί του θέματος. Για το θέμα τώρα της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Εξωτερικής Δράσης δεν έχω πρόβλημα με την ε, αλλαγή από προσωρινές σε μόνιμες θέσεις αλλά έχω πρόβλημα με το πρόγραμμα οργάνωσης ε, για τους υψηλόβαθμούς υπαλλήλους. Δεν μου δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για αυτή την αναδιάρθρωση και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν λόγοι να γίνει ανακατανομή του προσωπικού όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Αρχή Εξωτερική Δράση. Αυτό που ε, κατανοώ είναι ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι νέος οργανισμός ο οποίος ακόμα οργανώνεται και θα πρέπει να προσαρμόσει τον προγραμματισμό του καταλήλως. Αλλά αυτό δεν επαρκεί για να δικαιολογεί τον τόσο σημαντικό βαθμό αλλαγή θέσεων από θέσεις μεσαίας στάθμη σε υψηλόβαθμες θέσεις η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα για το προπολογισμό του 2012. Το Συμβούλιο έχει αποκρισταλώσει τη θέση του και έχει προσαρμόσει το προπολογισμό όσο προτάθηκε. Εγώ πρέπει να πω ότι με εκπλήσει αυτό, διότι στι άλλε περιπτώσει, το Συμβούλιο είχε πολύ αυστηρή θέση και προσπαθούσε να εξοικονομήσει χρήματα όπου μπορούσε. Και επομένω δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική διέπει αφενό ε, τη μείωση τη επισητιστική βοήθεια για του φτωχότερου Ευρωπαίου και από την άλλη ε, επιτρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες υψηλόβαθμες θέσεις για τους ε, υπαλλήλους των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων. Πρέπει φυσικά να είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε εδώ και μία επιλογή θα ήταν η Ευρωπαϊκή Αρχή Εξωτερικής Δράσης να αποκλείσει στους υπολογισμούς του το 1 τρίτο του προσωπικού το οποίο θα πρέπει να προέλθει από τα κράτη-μέλη και θα είναι αποσπασμένοι εμπειρογνώμονε. Έτσι θα μειωθεί ο αριθμό των υψηλόβαθμων υπαλλήλων που ζητούν τα κράτη-μέλη για την αρχή αυτή. Τέλος, επειδή η πρότασή μου σας απεστάλλει ε, καθυστερημένα, προτείνω να ε, αναβάλουμε την ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στις 12, αν συμφωνείτε. Πολύ σαφής η πρόταση, ο κύριος Βόκεν ε, έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις ανησυχίες και νομίζω ότι απεστάληκε σχετικό email από τον συνάδελφο, από τον κύριο Καλτιέρη, για τις ανησυχίες του και μάλιστα λέει ότι διασκεδάστηκαν οι ανησυχίες του από την κυρία Τρούπελ Νομίζω ότι η βασική του ανησυχία ήταν το, η κατανομή ενό τρίτου, δύο τρίτων. Τα δύο τρίτα να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι υπόλοιποι από τα κράτη-μέλη. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια κάποιε ακόμα ανησυχίε, όπω μα είπε και η συγγήτρια, και, συμφωνίζουμε και ε, συμφωνούμε συγγνώμη, και εμεί για την αναβολή τη ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Καλώ. Όντω φαίνεται λογική η πρόταση. Μετά τα επιχειρήματα που ακούσαμε και από την εισηγητριά μα Και αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει προτείνω να παρατείνουμε για τις 27 Σεπτεμβρίου για μία εβδομάδα δηλαδή την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες ώστε να διαμορφώσουμε καλύτερα τη θέση μας ε, ακούγοντας τις σοβαρές επιφυλάξεις ηγήτριας επί των αρχικών προτάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Alors, nous Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, θα ήθελα τώρα να αποταθώ στον Γκέραν Φέρμ, που είναι ο εισηγητής μας για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Μάλιστα είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα του δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει για την πορεία των συζητήσεων. Σας ευχαριστώ όπως βλέπετε έχει υποβληθεί το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από κοινού από τους ηγητές που είναι αρμόδιοι για την Ανατολική και την Νότια Γειτονία και αφορά την αναθεώρηση της, του Μηχανισμού Πολιτικής Γειτονίας και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον. Περίπλοκο το θέμα της πολιτικής γειτονίας γιατί έχει κάποια ευαίσθητα σημεία που τα αντιμετωπίσαμε και με τις μεταφορές του 2011. Θα επαναληφθούν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2012, αλλά η αναθεώρηση είναι τέτοιες εμβέλειες που μας υποχρεώνει να θετήσουμε πιο μακροπρόθεσμη άποψη. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών φυσικά θέλει να ε, επιμείνει στα δημοσιονομικά σκέλη της αναθεώρησης, αλλά υπάρχουν και πολιτικά τα οποία αφορούν περισσότερο την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Πάντως διαπιστώνουμε στην πρώτη παράγραφο της γνωμοδότησής μας ότι η πολιτική γειτονία μας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται μόνος ε, βοήθεια. Είναι σημαντική η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μια πτυχή οικονομικής ολοκλήρωσης που επίσης είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή τη διάσταση. Στη δεύτερη και την τέταρτη παράγραφο αναφερόμαστε στην περίπλοκη περιλυσύνθετη φύση των διαφόρων προτάσεων που υπευλήθησαν, το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Ιουνίου είπε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με τις μακροπρόθεσμες πτυχές, το ρόλο δηλαδή του μηχανισμού γειτονία στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως το σημαντικό είναι αυτά που λέμε τώρα να υποβληθούν και σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τι έγιναν ε, και στην, ε, στον προπολογισμό του 2011-2012 υπό βραχυπρόθεσμη άποψη δηλαδή, αλλά να έχουμε υπόψη και το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη πτυχή. Είχαμε κρίσιμες καταστάσεις στη νότια της Μεσογείου, στη Βόρεια Αφρική και για πολλά χρόνια αφιερώσαμε πολλά κονδύλια και στο ισχύον ε, μηχανισμό ΜΕΝΤΑ και στο συνεχίζονται και στο προηγούμενο. Ποια ήταν τα αποτελέσματα όμως αυτής της βοήθειας και αυτών των κονδυλίων. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ε, υποστηρίζαμε τη, τη διαμόρφωση δημοκρατικών θεσμών και ίσως τελικά διαπιστώσουμε ότι ενισχύαμε δικτατοριακά καθεστώτα. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Επίσης υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά σημεία, αλλά υπάρχουν και θέματα διαμόρφωση δημοκρατικών θεσμών, πολιτικά κτλ. Είμαστε αρκετά λοιπόν απαιτητικοί και κριτικοί σε αυτά που κάνουμε, ώστε να βελτιώσουμε τα μελλοντικά μας μέσα. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε και ένα συντονισμό των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα φτάνουν από τον υπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχουμε και σημαντικές ενισχύσεις από την ΕΤΕ, από την ΠΕΡΤ κτλ. Για να αξιοποιήσουμε λοιπόν τα κονδύλια στο έπαρκλο θα πρέπει να συντονιστούμε ώστε να αποφύγουμε επικαλύψεις και επαναλήψεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Επισημαίνουμε και το κίνδυνο να επικεντρωθούμε μόνο στην Αραβική Άνοιξη, στα γεγονότα στη Λιβύη, την Ισία, Αίγυπτο. Αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα και στην Παλαιστίνη, που επίση εμπίπτει στο μηχανισμό ε, γειτονία και τη χρηματοδότηση τη Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και το πρόεδρο Ούνερα των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ανέκαθεν τη γνώμη ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ επιφυλακτική πολιτική για να μην πω κοντόφθαλμη ώστε κάθε χρόνο στο σχέδιο προπολογισμού να μειώνονται σημαντικά τα κονδύλια για την Παλαιστίνη. Και αυτό το έκανε με πολιτικές προθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασκήσει πίεση σε άλλους δωρητές, αραβικές χώρες κυρίως. Φοβούμε όμως ότι αυτή η τακτική είναι αναποτελεσματική. Γιατί πραγματικά μας περιορίζει σε πολύ κοντόφθαλμη προσέγγιση της Παλαιστινιακή ε, Αρχής και των προγραμμάτων τη Σούνερα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και εδώ πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση και προοπτική. Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα είναι η ισορροπία μεταξύ Ανατολή και Νότου. Είχαμε πει ε, ένα τρίτο ανατολικά, δύο τρίτα για τον Νότο. Αυτή ήταν η κατά παράδοση αναλογία, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε άκαμπτοι να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις, ε, στις, ε, στα γεγονότα, στο δυναμικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη διάσκεψη Euronest στο Στρασβούργο και οι χώρες Ανατολικής Γειτονίας ε, δείχνουν μια ανησυχία για την υπερβολική προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότο. Και η Ανατολική Γειτονία μας είναι σημαντική για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί πολύ πιθανό στο μέλλον κάποια μέλη της Ανατολικής Γειτονίας ίσως ε, γίνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον συσφίξουν τις σχέσεις πολύ περισσότερο και συνδεθούν πολύ πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό να το λάβουμε υπόψη ότι αφορά την ισορροπία μεταξύ της γειτονίας προς Ανατολάς και προς Νότο. Προτείνουμε επίσης ε, ε, τις δυνατότητες εγγενείων προγραμμάτων και οργανισμών ευρωπαϊκών στις χώρες αυτές και μιλήσαμε και για το συντονισμό. Ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι ότι έχουμε πληθώρα προτάσεων για νέους μηχανισμούς. Βοήθεια για την Αραβική Άνοιξη, επιπαντός επιστητού, για την οικονομία, τη γεωργία, περιφερειακή πολιτική, δημοκρατία, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, σωρία προτάσεων, αλλά προσοχή προσοχή όλες οι δράσεις μας ε, να είναι καλά χρηματοδοτημένες, να αξιοποιηθούν και να συνοδευτούν από αιρεσιμότητα ώστε πραγματικά να αξιοποιηθούν σωστά τα κοινοτικά κονδύλια. Η παράγραφος 10 είναι από τις πιο επίμαχες γιατί το 1 πέμπτο του προγράμματος κανονικά θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και αυτή η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε ε, τέτοια κονδύλια από την ΕΤΕ ε, βρήκε αντίθετα πολλά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και αποτελματώθηκε. Πάντω ε, η Επιτροπή επιμένει ότι το 1 πέμπτο θα πρέπει να χρηματοδοθεί από reflows τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και αν δεν ε, αλλάξουν γνώμη τα κράτη-μέλη θα έχουμε μια τεράστια τρύπα στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ένα 20% μα λείπει. Θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να το λύσουμε. Και εμείς είμαστε υπέρ της χρήσης των reflows από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο συντονισμό μεταξύ Ένωση και κρατών μελών. Εμίζον πρόβλημα ανέκαθεν, ειδικά για την Βόρεια Αφρική. Πολλά κράτη-μέλη έχουν για τη Βόρεια Αφρική ιστορικούς δεσμούς, ε, συγκεκριμένες μεμονωμένες σχέσεις με μεμονωμένες χώρες, εξυπηρετώντας τα εθνικά του συμφέροντα, Ιταλία στη Λιβύη, Γαλλία στην Τινησία και ούτω καθεξής και πραγματικά υπήρξε αισθητή έλλειψη συντονισμού μεταξύ των μεμονωμένων χωρών μελών και των δράσεών τους στην ε, Βόρεια Αφρική και των κοινοτικών δράσεων. Από αυτήν την άποψη χρειαζόμαστε, παραλαμβάνω, καλύτερο συντονισμό και για πολιτικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους και το σημαντικό είναι όλες οι αιτήσει που έγιναν και εκλείσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να γίνουν ακουστές. Έχουμε ένα ιστορικό βέβαια πολλών μεγαλεπίβολων υποσχέσεων, αλλά που έμειναν ανεκπλήρωτες. Να μην επαναληφθεί αυτό και στην Αραβική Άνοιξη και στην πολιτική γειτονία. Αυτά ως προς την γνωμοδότησή μου και περιμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις των συναδέλφων. Η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 12 Οκτωβρίου, οπότε έχετε αρκετό χρόνο για να καταθέσετε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, Γιώραν. Ο κ. Χάρτουγκ. Σας ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα, όσα, από τα όσα άκουσα από τον κύριο Φάρμ. Θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια αυτοκριτική. Τα τελευταία χρόνια δόθηκαν πολλά χρήματα για υποστήριξη δικτατορικών καθεστώτων, κυρίως στη Βόρεια Αφρική. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος εν ώψη των ε, νέων δημοκρατικών εξελίξεων. Διερωτώ με όμως προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αυτές οι χώρες. Ακούμε από εδώ και από εκεί Αλαχού Ακμπάρ, ακούμε για Σαρία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν δίνουμε χρήματα για το πού θα πάνε και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Βεβαίω η επίγουσα ε, βοήθεια είναι ε, απαραίτητη, αλλά θα πρέπει η πρόοδος των χωρών αυτών να εξασφαλιστεί με τα δικά τους μέσα κυρίως. Βρίσκω πολύ δικαιολογημένη την ε, παρατήρησή σας κύριε συνάδελφε, απάντηση του Πρόεδρου. Ή αν έχει ζητήσει το λόγο, Γένσεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώραν Θάρμ για την εξαιρετικά διαυγή παρουσίαση του θέματος, καθώς και για την εξαιρετική εκθεσή του. Η ομάδα μου υποστηρίζει την ε, προσέγγιση του. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα το κείμενό του. Βρίσκω όμως ότι η προσέγγιση είναι πολύ ισορροπημένη ο κ. Χάρτονγκ είπε ότι ίσως να μην εύκολο, να μην αποδειχθεί εύκολο να υποστηρίξουμε την Αραβική Άνοιξη, αλλά ποτέ δεν ήταν και εύκολο να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές. Θυμούμε το European Training Foundation, το, ίδρυμα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου όταν προσπάθησε να συνεργαστεί με τις Αιγυπτιακές αρχές, χρειάστηκε να συνεργαστεί με 22 διαφορετικά υπουργεία και χρειάστηκε να αναπτύξουν πάρα πολύ ε, ευέλικτες τεχνικές ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν με τους νέους της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλές προθέσεις κατ' επανάληψη και το έχουμε αποδείξει αυτό όσο μπορέσαμε, ε, δοθισών των συνθήκων, αλλά ίσως οι συνθήκες αυτές να είναι και δύσκολες και στο μέλλον. Ο Γιώργαν έχει δίκιο που λέει ωστόσο ότι οι πολιτικές γειτονίας έχουν πολλές πτυχές και συχνά αναφέρονται σε θέματα τεράστιου ενδιαφέροντος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια έχει δίκιο όταν λέει ότι χρειαζόμαστε καλύτερο έλεγχο του, της βοήθειας προς την Παλαιστίνη. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα και όχι μόνο μια περιπτωσιολογική προσέγγιση και η πολιτική αστάθεια που παρατηρείται είναι επειδή λείπει ένα καλό ε, προγραμματικό πλαίσιο. Υποστηρίζω λοιπόν εν τέλει την έκθεση του Γιώραν. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αστερνίζομαι σε μεγάλο βαθμό τις παρατηρήσεις του κύριου Φάρμ, ιδιαίτερα τα σχόλιά του για την Παλαιστίνη συμφωνώ απόλυτα και με την κυρία Γέννησεν σε ό,τι αφορά την Αραβική Άνοιξη έχω κάποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις. Καταρχήν, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η αύξηση των πιστώσεων για την βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία στην Μεσόγειο να μην γίνουν ε, σε βάρος ε, της ε, υπόλοιπης Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Να μην βγάλουμε δηλαδή από τα κονδύλια της Λατινικής Αμερικής της υπόλοιπης Αφρικής για να ενισχύσουμε την Αραβική Άνοιξη. Προσοχή στην εξορρόπηση των κονδυλίων για τη συνεργασία. Δεύτερη μου ανησυχία. Σχέση ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών. Κατά κανόνα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, η αναλήψη υποχρεώσεων υπάγονται ε, ή ε, εκπορεύονται από συμβάσεις που εξετάζονται από, τη, από τα κοινοβούλια των χωρών που είναι αποδέκτες αυτών των συμβάσεων. Όταν όμως έχουμε μία περίπτωση άνοιξης ήδη το φθινόπωρο, με προβλεπόμενες εκλογές για τα τέλη του τρέχοντος και τις αρχές του επόμενου έτους, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός όπου όλες οι διαδικασίες να περάσουν από τις συμβάσεις ε, ε, αυτών των το μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των ε, νέων δημοκρατικών χωρών ίσως δημιουργηθεί μία ρήξη σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα σύναψη συμβάσεων και να δημιουργηθεί ακόμη ένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ ανάλυσης υποχρεώσεων και πληρωμών. Αυτό να το αποφύγουμε θα προτιμούσα. Και τέλος, πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά χρόνια συντήρησε απολυταρχικά καθεστώτα. Βέβαια, σε αντίθεση με την Τινησία, η Αίγυπτος ε, απορρίπτει την παρουσία διεθνών παρατηρητών στις επόμενες εκλογές. Και μάλιστα στα πλαίσια ενός εκλογικού συστήματος, όπου η μισή βουλή ε, εκλέγεται στον πρώτο γύρο με ένα ιδιαίτερο σύστημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μήπως, ε, να συζητήσουμε μήπως η Αραβική Άνοιξη γίνεται όμοιρος ε, ενός στρατιωτικού συστήματος ε, που προστατεύεται κυρίως από τους μουσουλμάνους, μάλλον ακραίους μουσουλμάνους, η Συντόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γκέραν για την πολύ καλή του γνωμοδότηση, πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης που πραγματικά επισημαίνει πολύ εύστοχα τα πιο σημαντικά θέματα και κυρίως τις δημοσιονομικές πτυχές της αναθεώρησης της πολιτικής γειτονίας. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να εμπλακούμε εδώ συζητήσεις που κανονικά αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Εγώ θα επικεντρωθώ σε δημοσιονομικές μόνο Αυτό που μου άρεσε στις προτάσεις σου, είναι ότι ε, αντιλαμβάνεσαι και εσύ την ε, όθηση αυτή που δίνεται με την Αραβική Άνοιξη και πιστεύει ότι το έργο μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η κατάλληλη στιγμή και η συγκυρία για την αναθεώρηση της χρηματοδότησης της πολιτικής γειτονίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δύο μόνο συγκεκριμένες παρατηρήσεις έχω για κάτι που κατά τη γνώμη μου θα συζητηθεί περισσότερο στο μέλλον. Αφορά τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση της ε, Παλαιστινιακής Αρχής. Τον προγραμματισμό της βοήθειας και τη χρηματοδότηση που θα στείλουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή. Εμείς είμαστε πάντα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την προσημείωση κονδυλίων για συγκεκριμένα εδάφη, συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένους δικαιούχους. Αυτό πάντα είναι επίμαχο θέμα. Αλλά ιδιαίτερα προβληματικό θα γίνει αν αυτή η προσημείωση γίνει με το συγκεκριμένο μηχανισμό. Αν παρεστεί ανάγκη, και φαντάζομαι θα μας επισημάνει η Ευρωπαϊκή ΑΦΕΤ αυτή την προσημείωση των κονδυλίων, ίσως θα πρέπει να τα αποσύρουμε από το νέο μηχανισμό Ανατολικής Γειτονίας. Πάντως με την παρούσα μορφή είναι αρκετά προβληματική κατά τη γνώμη κατάσταση. Ένα σχόλιο που δεν είναι και πολύ δημοσιονομικό, αλλά φαντάζομαι δεν θα σας εκπλήξει, ξέρετε ότι είμαι Πολωνέζα. μα ανησυχεί, με ανησυχεί ιδιαίτερα η απόσπαση τη προσοχή από χώρε όπω η Ουκρανία και η Λευκορωσία και ο προσανατολισμό αλλού, γιατί και η Ουκρανία και η Λευκορωσία έχουν πολύ σημαντικά θέματα, προβλήματα, ακόμη και ε, με τη δημοκρατία την, την ίδια. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Και πραγματικά θα με ενοχλούσε η επικέντρωσή μα στην Αραβική Άνοιξη να γίνει βάρος τη προσοχή μας προς την Λευκορωσία και την Ουκρανία, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και μάλιστα οξύνονται και όλα τα προβλήματα αυτά. Και χαίρομαι που μιλήσατε για μια ε, κριτική αναθεώρηση των προγραμμάτων μας για την κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία για να δούμε πραγματικά αν είναι σωστά προσανατολισμένα τα προγράμματα και πραγματικά περιλαμβάνουν και μια αξιολόγηση της, προέδρου, της πρόοδου και αν πραγματικά συνδυάζουμε την, ή εξαρτούμε την παροχή βοήθειας με τον πραγματικό εκδημοκρατισμό της χώρας δικαιούχου. Πολύ σωστή πρόταση και νομίζω ότι η γενική επισκόπηση που κάνει στον προβλημάτων είναι πολύ εύστοχη. Ευχαριστώ, Συντονία. Ο κύριος Αλφόνση. Euh, euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους σοσιαλιστές και τον εισηγητή μας, τον κύριο Φάρμ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συζήτηση επί της ουσίας για τα θέματα αυτά, γιατί το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη γειτονία της σε μεγάλο βαθμό. Είτε αν μιλούμε για διεύρυνση, γιατί και για τα Βαλκάνια δεν μιλούμε βέβαια, αλλά είναι σημαντική περιοχή. Και όσο εξελίσσονται τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι η αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου στι γειτονικέ μα χώρε θα αποτελέσει αναπτυξιακό παράγοντα και για την Ευρώπη και τι επιχειρήσει και τα προϊόντα τη. Ουσιαστικά αυτό είναι επένδυση στο μέλλον μα αυτή η επιδίωξη βελτίωση τη πολιτική γειτονία μα. Η ομάδα μου είναι υπέρ τη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και τη αναδιοργάνωσης αυτής της πολιτικής. Να μην ξεχνούμε φυσικά τα Βαλκάνια, να μην ξεχνούμε την Ανατολή, αλλά να είμαστε προσεκτικοί και ως προς εξελίξεις ε, στην Μεσόγειο, γιατί υπάρχουν πολλά διακυβευόμενα και ως προς τη μετανάστευση και ως προς το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική η γνωμοδότηση ζητά ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Εμείς είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι από τον εισηγητή, γιατί θεωρούμε ότι όσο πιο πολύ επίπεδη είναι η συνεργασία μεταξύ πόλεων και περιφερειών, τόσο πιο απτές ε, είναι οι πρόοδοι για το μέλλον της δημοκρατίας και της ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Και καλό θα είναι η γνωμοδότηση να περιλάβει και το ρόλο των μακροπεριφερειακών πολιτικών στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Μπόκρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία τεχνική παρατήρηση. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω την πολιτική συζήτηση παρά το γεγονός ότι και εγώ έχω απόψεις επί του θέματος. Υπάρχουν διάφορες μορφές ενισχύσεων, υποστήριξης και αναπτυξιακής βοήθειας, οι οποίες έχουν και αντίστοιχες δημοσιονομικές συνέπειες. Αυτή η δημοσιονομική γραμμή που λέει ε, αξιολόγηση των επανεισρεών δεν μπορεί να γίνει και να επαναπρογραμματιστεί με τον ίδιο τρόπο με την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόκειται για επενδύσει. Αυτό θέλουμε στην ε, περιοχή. Αλλά οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν επί τη βάση των κερδών. Παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αναπτυξιακή τράπεζα, επομένω λαμβάνει υπόψη και κάποιε πτυχέ πολιτικέ ε, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν ε, ε, και επιπτώσεις ε, στα κέρδη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός ο οποίος θα πρέπει να δείξει ότι οποιαδήποτε επένδυση κάνει έχει και το αντίστοιχο κέρδος, την αντίστοιχη επιστροφή. Επομένως, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή η διαφορά αυτή και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ίδια γραμμή με τις προσημειωμένες πιστώσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσημείωση κονδυλίων για επενδύσεις οι οποίες ε, θα υποστηρίξουν άλλες μορφές επενδύσεων. Συμφωνώ λοιπόν ότι όπως είπαν και κάποιοι άλλοι, αυτή η γραμμή θα πρέπει να τη χάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς ε, τα όσα λένε κάποιες κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μια υποσημείωση ή κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να λέμε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεπενδυθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προς τις ίδιες χώρες, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης. λίγα σχόλια εκ μέρους μου. Όπως εξήγησε και ο Γιώραν, βρισκόμαστε σε περίοδο ταχυτάτων εξελίξεων στην περιφέρειά μας και προς Νότον και προς Ανατολάς. Σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί διάσκεψη κορυφής της ε, Ανατολικής εταιρική σχέση. Αύριο η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ίσω ψηφίσει για το θέμα τη ε, Παλαιστίνη. Επίσης μιλήσατε ορισμένοι εξημών για τη Λιβύη, την Αίγυπτο κλπ. Πράγματι λοιπόν είναι καλή στιγμή να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε για την αναγκαία προσαρμογή των μηχανισμών μας. Εξάλλου ας μην το εξή. Πρώτον, είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπως είπε και η Σουδανία, δεν είμαστε η Επιτροπή Εξωτερικών. Οι συστάσεις λοιπόν για τις πολιτικές επιλογές θα πρέπει να προέλθουν από την Επιτροπή Εξωτερικών πρωτίστως όλοι βεβαίως είμαστε πολιτικοί έχουμε απόψεις και τις εκφράζουμε και εδώ βεβαίως με την ψήφο μας αλλά οι αξιολογήσεις καθαρά πολιτικές θα πρέπει πρωτίστως να γίνουν από την Επιτροπή Εξωτερικών Τώρα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα έχει και αυτή σημαντικό ρόλο να παίξει, κυρίως από δύο απόψεις. αφενός γενικά τα όσα συμβαίνουν στις αραβικές χώρες ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια πραγματική γνήσια αυθεντική ευρωπαϊκή παρέμβαση για να γυρίσει σελίδα από κάποιες ε, πολιτικές βοήθειες που είχαν ε, που είχαν κάποιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, παρόλα αυτά είχαν και κάποιο απεικιοκρατικό χαρακτήρα. Και προσέχω τα λόγια μου διότι και εγώ προέρχομαι από μια χώρα με απεικιοκρατικό παρελθόν. Από τη στιγμή που ο νότος της ε, Μεσογείου, χώρες αφρικανικές που παλαιότερα ετέλεσαν υπό την κυριαρχία της ΑΒ Ευρωπαϊκής χώρας, αποκτούν τώρα δημοκρατικά καθεστώτα ελεύθερα που θα μπορέσουν να αποτελέσουν ισότιμους εταίρους απέναντί μας από κάθε άποψη θα έρθει τότε η στιγμή της Ευρώπης και η Ευρώπη πρέπει να πάρει τη σκητάλη μέσα σε ένα πνεύμα του 21ου αιώνα και όχι βέβαια μέσα στα πλαίσια του πνεύματος του 19ου ή του 20ου. Η Επιτροπή μας των Προϋπολογισμών τότε θα έχει κέριο ρόλο να παίξει από δύο απόψεις. Να διασφαλίσει ότι οι βοήθειες που ε, θα δίνουμε θα είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές οικονομικά, το ζήτημα δεν είναι να δαπανίσουμε το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και στον τομέα αυτό έχουμε πράγματι επαρκή πείρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των ε, μειονεκτουσών περιφερειών, βλέπετε τα μειοσυνοχής, στο εξωτερικό δε της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη γειτονία μας, οι διάφορες ε, ενισχύσεις προενταξιακές γειτονίας, ανάπτυξης άλλων ε, υπήρων και ούτω καθεξής. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία που μπορεί να μας δείξει ποιες είναι οι βοήθειες εκείνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν και ποιες όχι. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά την ευθύνη μας, ο ρόλος της, της Επιτροπής μας θα είναι δύσκολος. Θα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές. αμέσως μετά με την έκθεση της κ. Μπαλζάνη θα δούμε πώς εμφανίζεται ο τίτλος 4 του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 με τις τροπολογίες που έχουν ήδη εγκριθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών που ξεπερνούμε έτσι τα 500 εκατομμύρια ευρώ από το κατόφλι της κατηγορίας και θα πρέπει να γίνει κάποια επιλογή και οι συστάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών θα ληφθούν υπόψη θα εξεταστούν προσεκτικά από την πλευρά μας αλλά όπως είναι και ο άχαρος ρόλος του Υπουργού Οικονομικών μιας κυβερνήσεως δικός μας είναι ο ρόλος αυτός, ο άχαρος ρόλος να πάρουμε το ψαλίδι. Κύριε Σιγητά, ποια είναι τα συμπεράσματά σας μετά από την ανταλλαγή απόψεων που μόλις ε, διεξήχθη. Σας ευχαριστώ. Πρώτα ορισμένα σχόλια σχετικά με τα όσα λέχθηκαν από τους συναδέλφους μας. Πρώτα για τον κύριο Χάρτονγκ που θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε διότι φοβείται ότι τα ε, καθεστώτα που θα ξεπηδήσουν θα έχουν ισλαμικό χαρακτήρα, ισλαμιστικό χαρακτήρα. Αυτό για μένα είναι επιχείρημα εκ του αντιθέτου. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, διότι αν όχι εμεί, τότε ποιοι. Τότε θα καταλάβουν το κενό οι δυνάμει εκείνε οι οποίε δεν ε, λαμβάνουν υπόψη ούτε τη δημοκρατική, δημοκρατική αιρεσιμότητα, ούτε τι ε, άλλε σχέσει με την περιοχή αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό το επιχείρημα αυτό. Δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε καθεστώτα, αλλά να ενισχύσουμε την δημιουργία δημοκρατικών συστημάτων και ε, οικονομιών που να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ευρύ πνεύμα όσον αφορά την υποστήριξη μη κρατικών οργανισμών ε, και άλλων ε, ε, οργανώσεων. Γένσεν και Πόρτα τόνισαν ότι υπάρχουν τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, τη λειτουργία των θεσμών που δεν έχουν ακόμα ε, αρκετά αναπτυχθεί. Για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με, τις, την ανάληψη υποχρώσεων. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να, να ζητηθεί μάλλον την Κομισιόν να απαντήσει. Έχουμε όμως την ε, ομάδα παρακολούθησης τη νότια Μεσογείου εδώ στο Κοινοβούλιο όπου διεξάγει ακροάσεις με συμμετοχή ε, εκπροσώπων. Είχαμε πάει πριν από λίγες μέρες και στην Τίνιδα στο Γραφείο Πληροφοριών της Ένωσης. Είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Βέβαια υπάρχουν ακόμα, ε, ε, κυρίως αυτό που απαιτείται τώρα είναι επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν θα έρθει η ώρα όμω θα πρέπει να φτιάξουμε νέε σχέσει με του θεσμού αυτού που θα ξεπηδήσουν και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο ε, θέμα που πρέπει να τεθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά δηλαδή την ε, ε, σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων κλπ. Για την Σιδονία θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό που είπατε όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας και του μέσου γειτονίας, αλλά όταν θα συζητήσουμε τον προπολογισμό του 2012 και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όταν μιλούμε για ισορροπία μεταξύ Ανατολών και Νότου, Ιστορικά υπήρξε πάντα αυτή η ισορροπία 2 τρίτα 1 τρίτο που ποτέ όμως δεν έλαβε επίσημο χαρακτήρα. Η φόρμουλα αυτή δεν υπάρχει εγγράφος πουθενά σε κανένα εγγραφό. Είναι μια γενική πολιτική πρόθεση. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό για μας να διατηρήσουμε κάποια εύλογη ισορροπία έτσι ώστε η πολιτική γειτονία να χέρει αξιοπιστία και προ Νότον και προ Ανατολά. Δεν επιτρέπεται να το διακινδυνεύσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Σχετικά με τον προγραμματισμό της ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής, θα πρέπει να εξετάσουμε όντως τα τεχνικά θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε αυτό χρησιμοποιήθηκε, ή μάλλον οι πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν για να ασκηθεί πολιτική πίεση σε άλλους δωρητές στις ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Έθνη, σε αραβικές χώρες, λέγοντας ότι δεν θα αυξήσουμε εμείς τις δεσμεύσεις μας μέχρι ότου τι αυξήσουν και οι άλλοι. Αυτό το παιχνίδι ωστόσο έχει αποβεί πάντοτε σε βάρο τη Παλαιστινικής Αρχή, τη Παλαιστίνης. Και δεν επιτρέπει στην Παλαιστινιακή Αρχή να προγραμματίσει σωστά τι δραστηριότητε τη. Το ίδιο και ισχύει και για την Ούνρα. Δεν γνωρίζουν οι αρχέ αυτέ αν θα μπορέσουν να πληρώσουν τον επόμενο μήνα του μισθού των δασκάλων. Και υπάρχουν χιλιάδε δάσκαλοι γιατί η Άνρα στην ουσία διεξάγει τι υποθέσει του κράτους, διοικεί το κράτο. Αλλά δεν γνωρίζουν ποτέ οι άνθρωποι τη λίγες εβδομάδες πριν αν θα έχουν λεφτά για να πληρώσουν τον κόσμο. Αυτό είναι παράλογο. Έστω και αν υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Να κατανοήσουμε ότι είναι η εργασία αυτή απαιτεί καλύτερο προγραμματισμό για την υποστήριξη της κοινωνία των πολιτών, μη κρατικών οργανισμών κλπ. Αυτό πάντοτε υπήρξε πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αφενός η Κομισιόν δεν θέλει να μπει στην βοήθεια πάρα πολύ μικρής κλίμακας κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Θέλει να ασχολείται με τα μεγάλα και εύκολο να διαχειριστούν πρόγραμμα. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή. Υπάρχουν οι μικρές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν επαρκή υποστήριξη. Έχει ασκηθεί πολλή κριτική κατά του μηχανισμού υποστήριξης της Κοινωνία των πολιτών, του ΙΠΑ, που δεν έχει μπορέσει να προσφέρει βοήθεια σε μικρές οργανώσεις. Και εδώ πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Είναι σημαντική η βοήθεια για τις δημοκρατικές οργανώσεις, βεβαίως να μπορούν να ελέγχονται με λογικό τρόπο. Αναφερθήκατε και στην διδημοποίηση, ο κύριος Αλφονσίν το είπε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό στην περίπτωση αυτή το ε, εργαλείο αυτό. Για τον κύριο Μπόκρος, για τα reflows της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, σύμφωνοι. Αλλά η πρόταση της Κομισιόν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα reflows της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας για να χρηματοδοτήσουμε το 1 πέμπτο του προγράμματος τις λεγόμενες επανεισροέ. Τα χρήματα υπάρχουν. Χρησιμοποίηση λοιπόν των επανεισρώων που βρίσκονται ήδη στους λογαριασμούς της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα έχουμε και το πρόσθετο 20% με χρήση του μηχανισμού ευελιξίας αλλά θα φτάσουμε σε ένα πρόβλημα για το 1 πέμπτο του συνολικού προγράμματος αν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύση γι' αυτό και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τις επανεισροές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυτό προτείνουν ορισμένε χώρε μέλη είναι οι επανεισροέ αυτέ να καταλήξουν στα ταμεία του πάλι. Αυτό είναι πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και στον, στη δική μα συζήτηση περί προπολογισμού για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα. Ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα έτσι, κάπω θα πρέπει να λυθεί, διότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε το 1 πέμπτο του προγράμματο επειδή Ορισμένες χώρες μέλη αντιτίθεται στην ιδέα της χρησιμοποίησης των επανεισρωών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα χρειαστεί λοιπόν τότε να κατατεθεί άλλη πρόταση. Νομίζω βεβαίως ότι είναι λογικά τα επιχειρήματα της Κομισιόν υπέρ των προτάσεών της και θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει 12 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι Έχουμε προγραμματίσει να ψηφίσουμε στις 7 Νοεμβρίου, η αφέτηση στις 14 και η γνωμοδότηση θα περάσει την δεύτερη ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ώστε να προσαρμόσουμε την τελική ψηφοφορία σε πιθανές εξελίξεις. Ευχαριστώ λοιπόν. Σημείο 13. Αναβάλλεται κατά αίτημα του εισηγητού. Το ίδιο και το 14. Σωστά, κυρία Βέρτμαν. Ζητήσατε κι εσείς αναβολή. Για το σημείο 15 να πούμε δύο λόγια. Ο εισηγητής μας, η Βάιλο Κάλφιν, απουσιάζει. Γιατί δραστηριοποιείται στη χώρα του αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα πολύ εντατικά. Και το ευχόμαστε καλό κουράγιο. Μου ανέθεσε λοιπόν ο κύριος Κάλφιν να σας ενημερώσω Πολλές φορές άλλωστε στο παρελθόν μας ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Έγιναν πολλές συναντήσεις στα πλαίσια τριμέρους διαλόγου σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγύησεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσική απόρρια λοιπόν της προηγούμενης συζήτηση που είχαμε μετά από παρατήρηση του κυρίου Μπόκρος. Τελικά σχεδόν φτάσαμε σε συμφωνία και το Συμβούλιο ενέκρινε, ε, οριστικοποίησε τη θέση του στις 20 Σεπτεμβρίου και για λόγους ε, διοριών από τις 26 Σεπτεμβρίου μόνο υποβάλλεται επίσημα το αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ισχύουσα διαδικασία εκπνέει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς στο Κοινοβούλιο εντάχει το κείμενο. Καταρχήν έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου η έκθεση, ώστε να υπογραφεί και να τεθεί σε ισχύ εμπρόθεσμα, καιρός πριν την λήξη της προθεσμίας. Και μάλιστα η γραμματεία εδώ μου επισημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει το θέμα στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου και όχι στη δεύτερη. Αυτά ενημερωτικά ώστε να είστε έτοιμοι για ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ήδη στην επόμενή μας συνεδρίαση που θα γίνει σε αρχές Οκτωβρίου, 6 Οκτωβρίου. Επί της ουσίας έχουμε ήδη δώσει την συμφωνία μας επί της αρχής. Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο εισηγητής μας. Οπότε πιστεύω θα έχει οριμάσει η κατάσταση και θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε σε 6 Οκτωβρίου. Θα ήθελα τώρα, μια και έχουμε στην αίθουσα και τον εισηγητή μας για την πολιτική και την, ε, πολιτική, και την εισηγητρία μας για την πολιτική εκείνη τον ε, Μόνικα Βλάδη και τον κύριο Μάνικα να μας κάνουν ε, μία σύντομη ενημέρωση για το θέμα που αφορά το κεφάλαιο 25 η Μόνικα πρώτα ε, μάλιστα συγγνώμη για, το σημείο 25 της ημερήσιας ένταξης, πολιτική κινήτων. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα είμαι πολύ λακωνική. Μην διαβάζετε το Κόμπου News, γιατί είναι ανακριβείς οι πληροφορίες που είδαμε εκεί. Έχει η κυβέρνηση του κράτους αυτού πληρώσει δύο χρόνια το μίστομα και τώρα σταματά. Δεν ξέρω λοιπόν τι να πω περισσότερο. Πολύ σύντομα ωστόσο πρόκειται για το Ινστιτούτο της Ισότιμης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών Institute for Gender Equality στα Αγγλικά ενημέρωσαν παρόλο που δεν είναι ε, υποχρεωτική η κοινοποίηση διότι είναι κάτω του ορίου η χρηματοδότησή του. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2012 έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν άνευ είναι βέβαια κάπως ε, καθυστερημένη τώρα στην αναζήτηση των νέων χώρων, διότι για δύο χρόνια ε, είχαν τη δυνατότητα να παραμένουν μέσα εκεί άνευ Τώρα ε, βιάζονται βέβαια, χρειάζονται 1200 τετραγωνικά μέτρα Στη Λιθουανία υπάρχουν διάφορες δυνατότητες, άρα δεν προβλέπω να είναι και τρομερό το κόστος. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, το λάβουμε υπόψη. Θα προχωρήσουν στη σύναψη συμβάσεως μισθώσεως για τους επόμενους 9 12 μήνες, αφού δεν το έπραξαν όταν έπρεπε. Δεν έχει όμως σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, οπότε νομίζω να το αποδραματοποιήσουμε. Η μόνη παράκληση που έχω προς την Κομισιόν εν προκειμένου είναι να τονίσει τους διαφόρους οργανισμούς όταν γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένες να εγκαταλείψουν σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ένα κτίριο, να αρχίζουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν να ασχοληθούν με τη μετακόμιση, διότι έχει συμβεί αυτό τρεις και τέσσερις φορές τελευταία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σωστό να τεθεί υπόψη των οργανισμών ότι με τον τρόπο αυτό πρέπει να διαχειρίζονται το θέμα στο μέλλον, διότι δεν είναι, ε, δεν είναι απαραίτητο τέλο πάντων να έχουμε την τελευταία στιγμή να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Κατά τα άλλα, νομίζω να το εγκρίνουμε. Ο Μάνκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη Μόνικα Ωστόσο υπάρχει κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν είμαστε αρκετά συστηματικοί. Το μίσθωμα εκπνέει το Δεκέμβριο και τον Σεπτέμβριο ε, επιλέχθηκαν τρία νέα κτίρια για τον Οργανισμό για την Ισότητα των Φόλων. Έχουμε λοιπόν μία νέα πρόταση που είναι ρεαλιστική. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός οίκος που θα στεγάζει και το ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ισότητα των Φύλων και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε και μία προσωρινή λύση για το Ινστιτούτο ε, για 12 μήνες τουλάχιστον και ο λόγο για τον οποίο σας λέω ότι δεν είμαστε συστηματικοί είναι γιατί θεωρώ ότι αν συμφωνήσουμε τώρα ότι θα μπορούσαν να συστεγάζονται οι οργανισμοί αυτοί, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση και νομίζω ότι η πρόταση που ακούσαμε θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλου. Ευχαριστώ. Η Μόνικα. Να προσθέσω ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι απολύτω αθώο και γι' αυτό η υπόδειξη αυτή θα πρέπει να γίνει και στο ίδιο το κοινοβούλιο, διότι εκεί έχει δίκιο ο κύριος Μάρκα, ε, συστεγάζονται τα όργανα εκεί και φαίνεται ότι και τα τρία δεν πρόσεξαν αυτή την καταληκτική ημερομηνία. Θα ήταν σωστό λοιπόν να, θα ήταν σωστό, λοιπόν, να αρχίσουν νωρίτερα να ψάχνουν για να βρουν και κάποια μισθώματα ευνοϊκότερα. Δεν είναι πάντω, όπως είπα και δραματικό διότι υπάρχουν αρκετοί χώροι. Δεν πρόκειται για το Παρίσι. Στο Παρίσι ήταν διαφορετικά και πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλώ. θα, συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια, με την έγκριση και του κύριου Μάνικα. Ήμασταν πολύ γρήγοροι σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχικά είχαμε προβλέψει συζήτηση και των τροπολογιών για τα σχέδια προϋπολογισμών του 2012 και για την Επιτροπή και για τα λοιπά τμήματα. Πρώτα οι συντονιστές και μετά ολόκληρη Επιτροπή το απόγευμα. Είναι όμως μόνο 11 παρά 20. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε τη συζήτηση τώρα. Να συνεχίσουμε με τους συντονιστές και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το απόγευμα για να κερδίσουμε και χρόνο. Κύριε Φερνάντες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το πρωί έλαβε χώρα μια σημαντική συνάντηση διαλλαγής με το Προεδρείο και το Προεδρείο κατέθεσε διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να περιλάβει και κάποια νέα στοιχεία που θα δούμε στο προπολογισμό του 2012 και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε με ακρίβεια κατά τη δημοσίευση του σχεδίου προπολογισμού. Για παράδειγμα, τις συνέπειες από την ε, ένταξη της Κροατίας και την άφηξη 18 νέων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να μας ενημερώσει, να μας πει τη γνώμη του και θα ρωτήσω και τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για τις προτάσεις τους και τις συμβαστικές λύσεις. Ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι πραγματικά πλησιάζουμε σε κατάληξη συμφωνία με το Προεδρείο και με τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Θα τολμούσα μάλιστα να αποκαλούσε ιστορική αυτή τη συμφωνία. Γιατί αν συγκρίνουμε ότι επιδέχεται σύγκριση μεταξύ του 2011 και του 2012, αν συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 2012 με αυτόν του 2011, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις έκτακτες δαπάνες ε, λόγω ένταξης Κροατίας και των 18 νέων ε, ευρωβουλευτών, έχουμε 0,8% ουσιαστικά διαφορά. Κάτι που προϋποθέτει και σημαντικές και ε, πραγματικές περικοπές. Σε ό,τι φορά την Κροατία και τα 8 νέα μέλη, τους 8 νέους ευρωβουλευτές, έχουμε 1,9 ενημέρωση. Κάτι που ανταποκρίνεται σε αρνητική ουσιαστικά ανάπτυξη, μια και ο πληθωρισμός ε, είναι 2,5%. Αλλά αν αφαιρέσουμε την Κροατία και τις συνέπειες της ένταξης Κροατίας, αν αφαιρέσουμε τις συνέπειες από τους 18 νέους ευρωβουλευτές και αν αφαιρέσουμε και τις συνέπειες από, τους, τις 300, 300 περίπου νέες θέσεις λόγω εφαρμογής ειδικής Λισαβόνας, η αύξηση ε, τελικά θα ήταν στάξη μόνο του 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με λιγότερα κονδύλια έχει περισσότερο έργο, κάνει πολύ περισσότερα γιατί έχουμε, περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες δράσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οικονομίες, να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε αναλάβει μια δέσμευση και δεν θέλουμε να υπαναχωρήσουμε. Αλλιώς, οι προβλέψεις ε, του Απριλίου, αν αμφισβητηθούν οι, αναλήψεις, οι, οι δεσμεύσεις μας, θα καταπέσουν. Οπότε, δεν έχει νόημα μια τέτοια διαφυσβήτηση, γιατί δεν θα προλάβουμε εγκαίρως να είμαστε έτοιμοι. Και μια και είναι δυσχερής και η οικονομική κατάσταση, θέλουμε τις επιπλέον αυτές οικονομίες, εξοικονομίες, χωρίς όμως να διακυβεύσουμε τις δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε απέναντι στη διοίκηση, γιατί η διοίκηση έδειξε ένα άνοιγμα για επιπλέον εξοικονόμηση και είπαμε τον Απρίλιο 2,3% και να λάβουμε υπόψη και την Κροατία. Άρα να λάβουμε υπόψη και τους νέους 18, 18 νέους ευρωβουλευτές. Ήταν συμφωνία δύσκολη τότε και χρειάστηκε να περικόψουμε 50 εκατομμύρια περίπου ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση του Προεδρείου. Τώρα θέλουμε επιπλέον 25 εκατομμύρια οικονομίες, εξοικονόμηση. Στην πράξη θα είναι 27 τα εκατομμύρια. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Από τα 25 εκατομμύρια έχουμε τα 21 εκατομμύρια για κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά θα συμβάλλουν στο, στην νομοθετική αριστεία. Θα εξοικονομήσουμε 10 εκατομμύρια στη διερμηνία, άρα η, η συνεδριάσεις θα κρατάνε από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, και α, ευρωβουλευτές όπως εγώ που είναι σε πολλές αποτροπές και συμπίπτουν οι διάφορες συνεδριάσεις, τότε θα φροντίσουμε να μην συμπίπτουν περισσότερες συνεδριάσεις και αυτό θα συμβάλλει στην νομοθετική αριστεία, αλλά εξοικονομήσεις θα κάνουμε και στις μεταφράσεις ε, και στα θέματα ολομέλειας για τις γραπτές ερωτήσεις και αυτές οι εξοικονομήσεις δεν θα πρέπει να ε, διαφυσβητήσουν ή να διακυβεύσουν τις ε, διάφορες αρχές της Ένωσης και φυσικά και την αρχή της πολυγλωσσίας. Γι' αυτό και υπάρχει δυνατότητα υποβολής ε, αιτήσεων για μεταφράσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα. Συμφωνούμε όλοι για επιπλέον ε, οικονομίες στα ταξίδια. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί και αυτό είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τις πολιτικές ομάδες. Προτάθηκε μείωση κατά 5% των ταξιδιών και επίσης υπάρχουν προτάσεις ε, για αποθεματικά και μάλιστα το σχέδιο των αποταμιεύσεων των εξοικονομήσεων που έχει υποβάλει το Προεδρείο αφορά όλα τα είδη ταξιδιών και αποστολών. Εγώ πρότεινα αυτό το αποθεματικό να είναι της τάξης του 15%. Έχουμε και τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε κάποια κονδύλια και στις δημοσιεύσεις, στην ενέργεια, όλα αυτά τα ζητήματα θα τα εξετάσουμε πιο διεξοδικά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Οι προτάσεις μας για τις εξοικονομίες αυτές θα πρέπει να είναι νομότυπες. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει συνένεση, μία εξοικονόμηση για τους μισθούς είναι αδιανόητη γιατί διακυβεύει το καταστατικό και άρα είναι απαράδεκτη, δεν είναι νομότυπη. Επίσης, κάτι που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου, το Προεδρείο δεν μπορεί να μειώσει. Για παράδειγμα, έχουμε τις γενικές δαπάνες. Το Προεδρείο δεν μπορεί να τις μειώσει, αλλά μπορεί να τις παγώσει αυτές τις γενικές δαπάνες το Προεδρείο μπορεί επίσης να κάνει μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή μόνο μέχρι το ποσοστό του πληθωρισμού. Τώρα υπάρχει μια νομική αμφιβολία το κατά πόσο εμείς μπορούμε να εμπλακούμε στα ποσά. Πάντως με ένα ψήφισμά μας μπορούμε να ζητήσουμε από το Προεδρείο να προβεί στο πάγωμα. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Το Προεδρείο να προτείνει από μόνο του αυτό το πάγωμα και έτσι θα επιληθεί το πρόβλημα. Πραγματικά χρειάζονται πολύ σημαντικές προσπάθειες και όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε είναι πολύ σημαντικές και είναι άνευ προηγουμένου αυτή η αύξηση μόνο του 0,8% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, στο προϋπολογισμό μας και έχουμε και τις επιπλέον δαπάνες που μας φτάνουν στο 1,9%, αλλά ακόμη και με το 1,9% πάλι αρνητική είναι η αύξηση του προπολογισμού, δεδομένου ότι ο ο, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός είναι 2,5%, άρα πολύ μεγαλύτερος από το 1,9%. Εγώ ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για όλα αυτά τα θέματα, γιατί το σε μια μεγάλη διαλλακτικότητα και ένα άνοιγμα στις διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε με την αύξηση του προϋπολογισμού μας για 0,8%. Και αυτό άλλωστε είναι και ένα μήνυμα προς τα έξω και απόδειξη ότι μπορούμε να καινοτομήσουμε και με λιγότερα κονδύλια μπορούμε να έχουμε περισσότερο έργο και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδης, και κύριος Βόν. Σήμερα το πρωί Νομίζω ότι ήμασταν πολύ επιτυχείς. Ε, οι σοσιαλιστές υποστήριξαν τη θέση του εισηγητή για να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, κάτι λιγότερο του 2%. Ε, προτάθηκε το 0,99% και 0,8% για την προσαρμογή λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε και αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα για να φτάσουμε στο 1,9% και νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη των σοσιαλιστών ότι και τα ίδια τα μέλη θα πρέπει να δείξουν ότι συνεισφέρουν ώστε να εξοικονομηθούν ε, κονδύλια. Ε, προτείνουμε μείωση των ταξιδιωτικών εξόδων ε, και μείωση του GAB και συμφωνούν ε, τα μέλη σε αυτά και νομίζω ότι οι σοσιαλιστές θα το υποστηρίξουν και υπάρχει συνένεση σε όλες τις ομάδες για το θέμα αυτό. Ο εισηγητής αναφέρθηκε και σε κάποια άλλα θέματα όπως η ενέργεια, αλλά νομίζω το βασικό είναι τα 21 εκατομμύρια που προτείνονται για τις υπηρεσίες διερμηνίας και μετάφρασης και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το πρέπει να το εξετάσουμε όλο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπο που εργάζεται το Κοινοβούλιο και τα μέλη θα πρέπει να κατανοήσουν, να δεχτούν ε, ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αν καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα 21 εκατομμύρια θα είναι πολύ σημαντικό. Κάτι ακόμα, ε, οι σοσιαλιστές θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να εξετάζουμε μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων για το 2012, αλλά θα πρέπει να καθορίσουμε και κάποιες αλλαγές μακροπρόθεσμα και γι' αυτό έχουμε καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, να δούμε τα ταξιδιωτικά έξοδα ε, και θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να μειωθούν αυτά περαιτέρω ολοκληρώνοντας ένα σημείο που δεν κάλεψε και ο εισηγητή, ο οίκο τη ευρωπαϊκή ιστορίας. Εμείς ως σοσιαλιστέ, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή με τη νομική βάση που έχουμε επιτρέπεται το Κοινοβούλιο να μισθώσει και να ε, πληρώνει το κτίριο για τον οίκο της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας μέχρι ένα σημείο και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση ε, υπάρχει και μία πρόταση να υπάρχει μία διπηρεσιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ε, δυνατό, αν μας το επιτρέπει η νομική βάση. Μία πρόταση είναι, δεν είναι βέβαιο κατά πόσα θα μπορέσουμε να τη δεχτούμε, αλλά το θέμα είναι ότι το καλό νέο σήμερα είναι ότι οδεύουμε προς μία συμφωνία στα όσα έχουμε συζητήσει. Αυτά πράγματι είναι καλά νέα. Ο κύριος Μποκός. Μποκρός. Να προσθέσω κι εγώ ένα καλό νέο, στα λοιπά καλά νέα, εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Συντηρητικών ε, υποστηρίζω κι εγώ τον εισηγητή και νομίζω ότι τα κονδύλια τα οποία μας έχει παρουσιάσει συνάδουν με τις ιδέες και τις προτάσεις ε, της ομάδος μας ιδίως ε, η συνολική αύξηση του 1,9% και χωρίς την Κροατία και τη ε, Λισαβόνα το 0,8 ή το 0,5 αν καταφέρουμε να το προχωρήσουμε και μέχρι εκεί. Θα ήθελα επίσης να πω εδώ ενώπιον της Ολομέλειας Επιτροπής Προϋπολογισμών ότι οι αλλαγές αυτές δεν γίνονται μόνο γιατί άλλαξε η οικονομική κατάσταση, αλλά γιατί είναι και το σωστό. Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τον Απρίλιο η αλλαγή και μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Βον δεν αναφερόμαστε εδώ σε ε, εξοικονόμηση μόνο για μία περίπτωση, αλλά μιλάμε για διαφορετικές ε, αλλαγές, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να εξοικονομούμε χρήματα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, ως προς τις λεπτομέρειες, συμφωνούμε με την εξοικονόμηση 10 συν 11 εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνίας και εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό που μας είπε ο Γενικός Γραμματέας όταν ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό σήμερα το πρωί. Μπορούμε να έχουμε πολυγλωσία πλήρως με σωστή χρήση των πόρων. Επομένως, καμία από αυτές τις οικονομίες δεν θα στερεί το δικαίωμα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνίας ε, στη γλώσσα τους. Ο Κλάους Βέλε είπε ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο δεξιοδική πρόταση. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να είναι κατόπιν ετήσεως. Διότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου προσφέρεται η υπηρεσία χωρίς ε, να τη χρησιμοποιεί κανείς στη σημερινή πρωινή συνεδρίαση άλλωστε ε, ήταν προφανές. Υπήρχαν τρεις πολύ καλοί Ούγγροι διερμηνείς, οι οποίοι παρούχαν διερμηνία και εγώ ήμουν ο μόνος Ούγγρος στην αίθουσα, δεν τους άκουσα σε καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε νόημα λοιπόν να υπάρχει διερμηνία από τα Ουγγρικά, όταν όλοι λίγο πολύ μιλούσαν μια κοινή γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για την... Ε, ε, τεκμηρίωση. Μου στέλνουν συνέχεια κείμενα στα ε, ουγγρικά και εγώ δεν τα διαβάζω ποτέ. Αν μπορούμε λοιπόν ε, να έχουμε κατόπιν ετήσεως ε, πρόσβαση σε έγγραφα, σε μετάφραση εγγράφων και αυτό θα μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα. Όσον αφορά τώρα την πρόταση του εισηγητή για τα ταξιδιωτικά έξοδα, το 5% περικοπή είναι το ελάχιστο που μπορούμε να περικόψουμε. Εμείς συμφωνήσαμε ότι θα μπορούσαμε ίσως να ε, χρησιμοποιήσουμε περισσότερα και να έχουμε ένα ποσό στο αποθεματικό. Για το πάγωμα συμφωνούμε επίσης. Συμφωνούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια περικοπή και, προς αυτή τη, και σε αυτή τη γραμμή. Και νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ τη συνένεση και θα μπορούσαμε να τα υποστηρίξουμε όλα όσα ακούσαμε. Ο Μιγγέλ Πόρτα. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, συμφωνώ με τις προβλεπόμενες εξοικονομήσεις στη διερμηνία και τη μετάφραση. Γιατί πραγματικά αυτές οι οικονομίες διαφυλάσσουν την πολυγλωσία σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αντιλαμβάνομαι ότι ο συνάδελφος Μποκρός προτιμάει να μιλεί την αγγλική. Εγώ θα είχα κάποια προβλήματα στα αγγλικά, γιατί δεν μιλάω τόσο άπτε στα γαλλικά όπως ο συνάδελφος Μπόκρος, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω γαλλικά. Αλλά παρόλα αυτά δεν, μπορώ, δεν θέλω να μιλήσω γαλλικά για πολιτικούς λόγους. Επίτηδε το κάνω, γιατί αν αρχίσουμε να αποποιούμαστε των μητρικών μας γλωσσών και των εθνικών γλωσσών, θα διατρέξουμε ένα σοβαρότατο κίνδυνο. Θα διακυβεύσουμε την πολυμορφία και τη λογική λειτουργία στο ίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων εν γέννη. Τούτου λεχθέντος, συμφωνώ απόλυτα ότι αν δεν χρειάζεται, αν δεν χρειάζεται τα ουγγρικά ή τα πορτογαλικά ή τα γαλλικά ή ακόμη και τα αγγλικά σε μια συνεδρίαση, ε, να μην χρησιμοποιηθούν. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίβαρο. Όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα ή που θα εξυπηρετήσει κάποιους άλλους, είναι απαραίτητο αυτό το δικαίωμα να διαφυλαχθεί στο ακέραιο. Για παράδειγμα, στη συνεδριάση των συντονιστών, εγώ δεν έχω πάντα πορτογαλικά, Μερικές φορές μιλάω μέχρι και αγγλικά. Και αυτός ο κίνδυνος, ε, εδώ ελοχεύει ένας πολιτικός κίνδυνος. Είναι λειτουργικό με ένα τέτοιο σύστημα, αλλά είναι κάπως διστραμμένο. Δεύτερον, αρχίζει να διαφαίνεται πιθανότητα συμφωνίας για τα ταξίδια και η πρόταση μείωση των ταξιδιών κατά 5% και η δημιουργία ενός αποθεματικού με 15% νομίζω ότι είναι μία πρόταση αξιόλογη. Αλλά προσοχή, μία τυφλή περικοπή οριζόντια 5% σε όλα τα ταξίδια δεν είναι λογική λύση, δεν είναι εύστοχη λύση. Και η πρόταση να βάλουμε στο αποθεματικό 15% περίπου δηλαδή 12 εκατομμύρια ευρώ θα είναι εύστοχη λύση και θα είναι έμπρακτη λύση μόνο αν το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλει μία σωστή πρόταση για, τις, για τους γενικούς κανόνες αλλά και τις εξαιρέσεις που θα μας επιτρέπουν τη, το ταξίδι σε business. Αλλιώς μια τυφλή πολιτική θα έχει ένα τίμημα. Για παράδειγμα, στις αποστολές των επίσημων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών θα μειωθεί ο αριθμός των ε, ευρωβουλευτών που θα ταξιδεύουν. Κάτι τέτοιο όμως αποβεί εις πολιτικής α, ε, ε, αντιπροσωπευτικότητας μιας αντιπροσωπείας. Είμαι κατά οποιοδήποτε επιδείνωσης αυτής της αντιπροσωπευτικότητας των αντιπροσωπιών μόνο και μόνο στο όνομα ή στο βωμό ενός τυφλού κριτηρίου μείωσης και οικονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατηγορία γενικές δαπάνες. Εμείς λαμβάνουμε περίπου 52.000 ε, ε, ευρώ το χρόνο για έξοδο παραστάσεως και γραμματιακά έξοδα. Δηλαδή περίπου 4.500 ευρώ το μήνα. Έξοδα παραστάσεως και γραμματιακά έξοδα. Αυτό το επίδομα δεν έχει καμία δικαιολόγηση. Είναι τελείως δυσανάλογο αυτό το επίδομα δεδομένης κατάστασης. Είναι ουσιαστικά ένας έμεσος μισθός αυτά τα 4,5 χιλιάρικα και χωρίς καμία δημοσιονομική επίπτωση κοινοτική είτε εθνική. Μόνο και μόνο επειδή χαρακτηρίζεται ως επίδομα. Πιστεύω ότι σε αυτό το κονδύλιο που χρησιμεύει για τηλεφωνικούς λογαριασμούς, για αγορά, ε, χαρτιού, iPad, για τους βοηθούς, αλλιώς αγοράζαμε κάθε μήνα ένα υπάτο κάθε βουλευτής. Αυτό το κονδύλιο κατά τη γνώμη μου είναι υπέρογκο για το είδος των πόρων που χρησιμοποιούμε. Και σε αυτό το κονδύλιο είναι που θα πρέπει να κάνουμε περικοπές. Εγώ μάλιστα πρότεινα περικοπή 25%. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό αυτό το ποσοστό για μερικούς συναδέλφους. Η αρχή της περικοπής όμως, σε τέτοιου είδους δαπάνες θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και από αυτή την άποψη η συμφωνία στο σημείο αυτό φαίνεται απίθανη. Εγώ πάντως θα επιμείνω σε αυτό το θέμα μέχρι τελικής πτώσεως. Γιατί αυτό είναι... Μια τέτοια περικοπή δίνει ένα μήνυμα στους συμπολίτε μας ότι εμείς ως Ευρωβουλευτές είμαστε διατεθειμένοι να περικόψουμε και δικά μας κονδύλια και επιδόματα Πολλό δε μάλλον που δεν δικαιολογούνται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις ούτε επηρεάζουν το, την ποιότητα του έργου μας. Και δεν έχει καθόλου δημαγωγικό χαρακτήρα μια τέτοια πρόταση. Αντίθετα, νομίζω ότι η υπευθυνότητα και η λιτότητα μας υποχρεώνει να αποδεχτούμε ότι οι, οι περικοπές δεν θα πρέπει να αγγίζουν μόνο τις, τους φτωχούς, τις μικρές και μεσαίες τάξεις της Ευρώπης, αλλά και τους ευρωβουλευτές που δεν έχουν πληγεί από τις πολιτικές λιτότητες ούτε και έχουν ευκαταφρώνει τους μισθούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και παραλαμβάνω τη συζήτηση αυτή θα την συνεχίσω και θα επιμείνω μέχρι τελικής πτώσης, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Πρώτα η Helga Trüppel. Ε, Γενικά, νομίζω ότι κατευθυνόμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να είμαστε οικονόμοι και να κάνουμε μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές οικονομίες αλλά και ταυτόχρονα και μια ανανέωση, μια χρήση καινοτομιών. Να βρούμε δηλαδή υπεύθυνου τρόπους να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους. Αντιδρώντας έτσι βέβαια στην παρούσα κρίση και τις πολιτικές λιτότητας αλλά ο κ. Μπόκρος ε, λέει σωστά ότι πρέπει να προχωρήσουμε και πέραν αυτού. Να δείξουμε δηλαδή ότι είμαστε πολύ υπεύθυνοι σε ό,τι αφορά την δαπάνηση των χρημάτων και μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα. Μία πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Φερνάντες. Μου αρέσει που έβαλε αυτό το offsetting για το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά βλέπω ότι το αντιστάθμισμα δηλαδή, την αντιστάθμιση για το ε, ε, διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά δεν βλέπω να περιλαμβάνονται πλέον τα σημεία τα σχετικά με την ΕΜΑΣ. Τώρα θα πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι είναι καλό να, επανοργανωθούν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ώστε να γίνονται από τη Δευτέρα το απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το βράδυ για να μην θα πανώνται παραπάνω χρήματα ειδικά τρίτες και τετάρτες της εβδομάδας επειδή πέφτει το βάρος κυρίως εκεί αλλά να γίνει μια καλύτερη κατανομή των συνεδριάσεων και νομίζω ότι θα έχουμε και την σύμφωνη γνώμη των βουλευτών επ' αυτού. Το Προεδριό φάνηκε πρόθυμο να κάνει προτάσεις εξοικονόμησης σχετικά με τις μεταφράσεις ή τις διερμηνίες πώς είναι η διαχείριση των μεταφράσεων στις συνεδριάσεις μας. Αφενός πρέπει να διατηρήσουμε την πολυγλωσία. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πολύ καλύτερες λύσεις μιας καλής διαχείρισης και έτσι μόνο όταν απαιτείται μετάφραση να χρησιμοποιείται και όταν δεν απαιτείται να μην γίνονται οι δαπάνες. Είναι δηλαδή και ζήτημα ορθής διαχείρισης και υπεύθυνη στάση απέναντι στον προπολογισμό μας. Γενικά λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια περικοπή της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Αυτό θα ήταν καλό. Για το γενικό επίδομα τώρα. Πρώτα θα πω ότι στην χώρα μου, τη Γερμανία, υπάρχει τώρα δικαστική απόφαση που δέχεται αυτό το γενικό επίδομα. Τώρα έρχομαι στην τροπολογία μας για το θέμα ότι θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να δείξουμε και κάποια προθυμία αυτοπεριορισμού και να προχωρήσουμε σε ένα πάγωμα. Αυτό νομίζω είναι το λογικό. Έρχομαι τώρα στο θέμα των δαπανών ταξιδιού. Όλα τα τελευταία χρόνια, και χωρίς να θέλω να είμαι ούτε δημαγωγός ούτε λαϊκίστρια, πάντοτε είπα ότι υπάρχουν τρόποι για σύντομες πτήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούμε εισιτήρια flex οικονομικά και όχι απαραίτητα business. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, για μακρινές πτήσεις ή για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας ή ε, είναι μεγάλης ηλικίας, τότε να είμαστε πιο εύκαμπτοι. Νομίζω πάντως ότι εδώ μπορούμε επίσης να κάνουμε κάποιες εξοικονομήσεις. Και το Προεδρείο μιλεί για μια εξοικονόμηση της τάξεως ε, του 5%. Άρα και εδώ νομίζω κινούμαστε στην ορθή κατεύθυνση. Και υποσχέθηκαν ότι θα αναζητήσουν τρόπους για να μειώσουν τις δαπάνες. Και αυτό λοιπόν με βρίσκει σύμφωνη. Ευρωπαϊκός οίκος ιστορίας τώρα. Αυτό που θέλω να διασαφίσω είναι διότι το Προεδρείο είπε πάλι ναι, υπάρχει μια νέα τροποποίηση, διότι την Άνοιξη φέτος βρέθηκε μια συμβαστική λύση. Υπάρχουν όμως πληροφορίες που έχουμε τώρα και δεν είχαμε τότε, Άρα αντιδρούμε στο ότι μέχρι τώρα δεν ήταν σαφή η νομική βάση. Τώρα το Προεδρείο ισχυρίζεται ότι υπάρχει νομική βάση για το κέντρο επισκεπτών. Αυτό που θέλω εγώ να γνωρίζω, διότι μέχρι τώρα δεν έχω δει το τελευταίο business plan και θέλω να είμαι βεβαία ότι θα διατηρήσουμε τον έλεγχο των δαπανών, του κόστους. Διότι γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει το νέο κτίριο, τι σημαίνουν νέα κτίρια και η κατανάλωση, η νέα κατανάλωση και πολύ φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε σκάνδαλα τα επόμενα χρόνια δεθήσεις τη καταστάσεω στην Ευρώπη. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το business plan λοιπόν, ποιο θα είναι το κόστος για το κτίριο, αλλά και, τα επακόλουθα, και το επακόλουθο κόστος. Να βάλουμε και την Κομισιόν μέσα. Νομίζω ότι είναι σωστό να είναι κοινή δαπάνη για το νέο αυτό έργο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι σαφή πριν να μπορέσουμε ως πολιτική ομάδα να πούμε εμείς ότι ε, είμαστε σύμφωνοι. Είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν θα θελήσει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ε, πρωτομών όλων των προέδρων της από, την, ε, από τις αρχές μέχρι και του κ. Μπαρόσο. Ο κύριος Άλβαρο. Κύριε Πρόεδρε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής που έγινε σήμερα το πρωί σε συνεργασία με το Προεδρείο κατέστησε σαφές ότι ναι μεν ίσως υπάρχουν και κάπως διαφορετικές αποχρώσεις απόψεων αλλά ότι γενικά στο σύνολό τους οι συνάδελφοι δέχονται τις προτάσεις του εισηγητού Φερνάντες για εξοικονομήσεις στον τομέα της διερμηνίας και της μετάφρασης. Συνολικά μαζί με το Προεδρείο το επιτύχαμε αυτό και το Προεδρείο βέβαια και είναι κατανοητό αυτό ζήτησε να μην παραμείνουμε στις περικοπές μονάχα στο δημοσιονομικό τμήμα αλλά να εξετάσουμε και ως Επιτροπή Προϋπολογισμών τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι ε, περικόπες αυτές. Θυμούμε ότι ρώτησα εάν υπάρχει συνένεση στο θέμα ότι η περικοπή των πόρων θα οδηγήσει και σε διαρθρωτικές αλλαγές στην εργασία των Επιτροπών ώστε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η υπηρεσία της διερμηνίας. Δεν υπήρξε ένσταση εκεί. Ακούγοντας τον κύριο Πόρτας μου φάνηκε ότι ξέφευγε λίγο από την πορεία αυτή, αλλά μετά από ορισμένου ελιγμούς επανήλθε. Και βέβαια το δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται στην μετρική του γλώσσα και να έχει στη διάθεσή του και έγγραφα στη μετρική του γλώσσα, καταρχήν θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα είδος αυτοματισμού. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχει ανάγκη, όπως είπε ο κ. Μπόκρος, ακόμα και αν δεν τα χρειάζεται, του διατίθεται ωστόσο και τα έγγραφα και η ε, διερμηνία. Αυτό νομίζω είναι κατασπατάληση ε, των ε, πόρων. Και νομίζω ότι εάν σημειώσουμε ότι ο στόχος μας είναι μια οικονομική χρήση των υπηρεσιών. Εφόσον δηλαδή γίνεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο να έχει στη διάθεσή του τα έγγραφα αλλά και την ε, διερμηνία, αυτό να μπορεί να συνεχίσει να προσφέρεται. Τα μέτρα εξοικονόμησης δεν αποτελούν μονόδρομο, βεβαίως πάντοτε κάποιες εξοικονομήσεις ε, επιφέρουν και αλλαγέ. Και ω μέλη τη επιτροπή Προπολογισμών έχουμε το χρέο όχι μόνο να περιορίσουμε τις ε, αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε το θέμα κατάλληλα και στους υπόλοιπου ε, συναδέλφους μας. Είναι αυτό πάντω ένα μέρος τη ευθύνη που φέρουν τα μέλη τη Επιτροπή ε, Προπολογισμών και ευχαριστώ Όλε και όλους τους συναδέλφους που ε, συνένεσαν σήμερα. Τα άλλα ανοιχτά θέματα είναι τα έξοδα ταξιδιού, η μισθή και ο Ευρωπαϊκός Οίκος Ιστορίας. Για αυτό το τελευταίο δεν είμαι μετοχός, σας το λέω ήδη καθαρά. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι θα προτιμούσα να γίνει συγχρηματοδότηση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου, διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, ωφεληθεί με ομάδες επισκεπτών κλπ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αδιαμφισβήτητο. Ταυτόχρονα είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής και στα πλαίσια των περαιτέρω συζητήσεων θα κάνει προτάσεις και για το γενικό τμήμα των δαπανών. Εγώ συμφωνώ να πούμε ότι το παγώνουμε, άρα ονομαστικά έχουμε και κάποια εξοικονόμηση γιατί βρισκόμαστε κάτω από τον πληθωρισμό. Έχω και κάποια συμπάθεια για τις προτάσεις του κ. Πόρτας. Ήδη προκαιρού είχα προτείνει σχετικά πράγματα. Η πρότασή του δηλαδή μείωση κατά 500 ευρώ του επιδόματος γραφείου που για τον έναν ή τον άλλο θα σημάνει ίσως μια εφημερίδα λιγότερη αλλά τα 500 ευρώ τον μήνα θα σημάνουν στο χρόνο 450 εκατομμύρια ευρώ. Ας το σκεφτούμε λοιπόν αυτό. Όσον αφορά τώρα τις δαπάνες των μισθών. Υπάρχει βέβαια ε, δυνατότητα να λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή το Προεδρείο ε, να λάβει την αποφασιστική αρμοδιότητα εφόσον πρόκειται για διαθεσμική συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών που παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του προϋπολογισμού θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο εφόσον προχωρήσουμε σε αυτή την εξοικονόμηση. θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο αυτό με επιτυχία, έτσι νομίζω. Σήμερα είχα την ευχαρίστηση να εκπροσωπήσω τον πρόεδρό μας στην συνεδρίαση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την επικοδομητική και πειθαρχημένη εργασία σήμερα το πρωί. Χαίρομαι που υπάρχει τέτοια δυνατότητα καλής συνεργασίας μέσα στην Ευρώπη ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που διατρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Άλβαρο γιατί πραγματικά συμμετείχε με τον εισηγητή και τους συναδέρφους στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων και ήταν πολύ αποτελεσματικό Τον συγχαίρω. Και όπως λέμε στον αθλητισμό, όταν μία ομάδα κερδίζει, δεν τροποποιούμε τη σύνθεσή της, ούτε και εδώ θα το κάνουμε. Λάζλο Σούριαν. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Σούριαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τις διάφορες απόψεις των συναδέλφων, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να πούμε ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές έκανε εξαιρετική δουλειά. πριν από κάποιε εβδομάδε τα προβλήματα του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ε, πολύ ακαθόδε ζήτημα και τώρα καταφέρνουμε να προχωράμε και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ κάποιες απόψεις όσον αφορά τις προτομές των επιτρόπων που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να έχουμε προτομή μόνο των εκλειπώντων. Για όσους είναι ζωή σας παρακαλώ ποτέ. Μα θέλουμε να τους κρατήσουμε όλους, λέει ο Πρόεδρος. Πραγματικά ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα εάν βελτιώσουμε, βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα. Τέλος πάντων, πέραν ε, των ε, αστείων, Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στο ότι δεν θα έχουμε μετάφραση χωρίς να υπάρχει αίτημα για μετάφραση. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και είναι σημαντικό. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες διερμηνίας τις συνεδριάσεις, δεν ε, αρκεί να εξετάζουμε μόνο εάν υπάρχει ε, διερμηνία σε όλες τις γλώσσες και αν απαιτείται από όλες τις γλώσσες. Ε, υπάρχουν και οι βοηθοί μας οι οποίοι κάθονται στα ε, ε, πίσω έδρανα και μπορεί να παρακολουθούν ακόμα και αν απουσιάζει το τακτικό μέλος ή μπορεί να αντικαθιστάται από το αναπληρωματικό μέλος ε, αυτό έγινε ας πούμε, στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι εδώ, αλλά κάποιος με αντικατέστασε και ε, επομένως υπήρχε εκπροσώπηση. Επίσης, η πλειονότητα των συνεδριάσεών μας ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και πολλοί παρακολουθούν τι συμβαίνει στις συνεδρίες από το γραφείο τους. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι γίνεται χρήση των διαφόρων γλωσσών ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά τη διερμηνία, λοιπόν, είμαι κατά ε, οποιασδήποτε αλλαγής ε, του παράντος κανονισμού. Ε, ίσα ίσα σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών διερμηνίας και όχι να περιοριστεί. Όσον αφορά τώρα τις ταξιδιωτικές δαπάνες, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί ε, στις αρχές μας και να σας αναφέρω μόνο μία. Κάθε μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ισότιμο με τους υπολείπους. Οποιαδήποτε διάκριση λοιπόν είναι αδύνατη. Ωραία είναι να λέμε από την πλευρά μας ότι εγώ είμαι πέρα από όλα τα ηλικιακά όρια, ε, εάν υπάρξει ένα όριο ηλικίας. Αλλά είμαι κατά, κατάφορα κατά οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίσης είναι αστείο να λέει κάποιος ότι αν προσκομίσει ιατρικό ε, πιστοποιητικό έχει επιπλέον δικαιώματα σε σχέση με κάποιον άλλον. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω προς τη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι αρχίζουμε να φτάνουμε σε μία λύση για αυτή την τόσο, επιτρέψτε μου, ε, στη συζήτηση, διότι ε, βιώνουμε καιρούς λιτότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δείξει κάτι ουσιαστικό και όχι μόνο επί πολλές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ, και νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος και όλων των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια καταρχήν στον Ζωζέ Μανουέλ και στον πρόεδρο Άλβαρο για το έργο τους. Μία ερώτηση πρώτα. Διάβασα με ενδιαφέρον την πρότασή σας ε, για περισσότερες μέρες συνεδριάσεων και μείωση της, ε, του κόστους διερμηνίας αλλά έτσι θα αυξηθεί μαζικά το per η ημερήσια αποζημίωση. Γιατί αν αντί για τέσσερι μέρε συνεδριάζουμε πέντε μέρε, ναι, με θα έχουμε περικοπέ στον προπολογισμό διερμηνία, αλλά θα έχουμε αύξηση στον προπολογισμό ημερήσεων αποζημιώσεων. Ε, κάνατε τη σύγκριση και είναι όντω οικονομική αυτή η λύση που προτείνεται. Συμφωνώ και στενίζομαι τι επιφυλάξει για τον οίκο τη ευρωπαϊκή ιστορία. Εγώ θα πρότεινα να διοργανώσουμε και δημόσια ακρόαση για να δούμε τι γίνεται με, τα, με τις δαπάνες επενδύσεων και τις δαπάνες λειτουργίας, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να δεχτούμε κάτι που δεν είναι σαν το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά κάτι που είναι σχετικά περιθωριακό στο δικό μας πλαίσιο εργασιών. Ένα έτοιμα. Έχουμε καμιά ιδέα ποια είναι η γνώμη των, 25, των 27 εθνικών κοινοβουλίων για το θέμα αυτό. Για να έχουμε και μία εικόνα για τη δική τους θέση. Βέβαια, αυτά είναι δικά μας θέματα. Θα τα ρυθμίσουμε εμείς και στηρίζονται σε δεοντολογικά κριτήρια. Αλλά σκόπιμο δεν είναι να ρίξουμε μια ματιά και τι συμβαίνει και αλλού, στα άλλα κοινοβούλια. Γιατί τα κράτη-μέλη μας υποβάλλουν διάφορες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό, να ρωτήσουμε στα δικά τους κοινοβούλια τι μέτρα λιτότητας λαμβάνουν. Και τέλος για τα ταξίδια. Εγώ στο κοινοβούλιο ε, έμενα πάντα κατάπληκτος για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο ε, το, στο οποίο βρίσκει κανείς τα ακριβότερα ταξίδια του κόσμου. Και αν κανείς αποταθεί στο ταξιδιωτικό αυτό πρακτορείο, που δεν είναι ιστορικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να είστε βέβαιος ότι θα πληρώσετε διπλάσια και τριπλάσια τιμή από το ίδιο ταξίδι αν το βρείτε μόνο σας στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε λοιπόν να, να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να κάνουμε καλύτερο έλεγχο του κόστους ε, του ταξιδιωτικού. Και έτσι να προβούμε σε κάποιες οικονομίες με πιο οικονομικές τιμές στα ταξίδια. Πιστεύω ότι έτσι θα κάνουμε πολύ μεγαλύτερες οικονομίες από το περιοριστικό 5% που προτείνεται. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε και ανα πάσα στιγμή. Και δεν νομίζω ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο κόπτεται να βρει ανταγωνιστικέ τιμέ ε, για του βουλευτέ, γιατί δεν είναι κανένα αντίβαρο. Νομίζω ότι αν προσέξουμε το πρόβλημα σε πολύ πρώτερο στάδιο, θα εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερα από ό,τι υποχρεώνοντα του ε, ε, πιο ηλικιωμένου βουλευτέ, του 60 να ταξιδεύουν οικόνομοι. Η πρότασή σας να δούμε την κατάσταση στα, διεθνικά Κοινοβούλια είναι πολύ εύστοχη. Να δούμε τι κάνουν και εκείνα. Κύριε Άλβαρο, εν συντομία, ζητήστε το λόγο για να απαντήσετε στον κύριο Ρικέ. Μια σύντομη απάντηση. Ρωτήσατε εάν έχει γίνει πλήρης υπολογισμός, εάν θα αυξηθούν οι μερίσεις αποζημιώσεις. Ομολογμένως δεν συζητήθηκε η ιδέα αυτή, διότι εφόσον κανείς είναι απόν, δεν λαμβάνει και μερίσια αποζημίωση. Άρα εάν μια μέρα αν είναι κανείς παρόν μία μέρα παραπάνω, θα, ε, θα πάρει και μία παραπάνω ε, ημέρηση αποζημίωση. Θα με εκπλήξει πάντως αν υπάρξει μεγάλη διαφορά. Εγώ νομίζω ότι η εργάσιμη εβδομάδα είναι τουλάχιστον από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Βέβαια ο καθένας θα αποφασίσει για τον εαυτό του, αλλά για την ώρα στην παρούσα κατάσταση δεν μου φαίνεται ευφιές να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την ημερήσια αποζημίωση. Ε, έχω μια ιδέα για το πώς θα τη η κοινή γνώμη τη συζήτηση αυτή ε, μέσα σε περίοδο κρίσεως. Ανεξαρτήτως τώρα του εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι λογικές αυτές συνέπειες, είναι διαφορετική η υπόθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τις ε, δαπάνες ταξιδιού, έχετε απόλυτα δίκιο. Και εμείς στην ομάδα εργασίας είδαμε ότι στο γραφείο ταξιδιών οι τιμέ είναι υψηλότερε από ό,τι συνήθω. Αλλά δεν υπάρχει και καθήκον, δεν υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κανείς το γραφείο ταξιδίων. Μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο καλύτερες τιμές. Ε, κύριε Μάνκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει πρόγραμμα συνεδριάσεων, Άλλε επιτροπές έχουν διαφορετικό πρόγραμμα συνεδριάσεων και δεν μεταφράζονται όλα τα έγγραφα σε όλες τις γλώσσες, πολλές φορές λόγω έλλειψη χρόνου η πάγια πρακτική είναι συνήθως να υποβάλλονται αυτές οι μεταφράσεις, κατόπιν εορτής βέβαια, οπότε είναι και άχρηστες για μας. Ίσως θα έπρεπε να λάβετε αυτό υπόψη και να εξοικονομήσουμε χρήματα σε αυτή την περίπτωση. Όταν ήμουν εισηγητής για το 2010 για τον προπολογισμό των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησα να παρακινήσω και τα υπόλοιπα μέλη να κάνουμε έναν έλεγχο για να παρακολουθήσουμε πώς συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όταν όταν έκανε το ελεγκτικό συνέδριο την αντίστοιχη διαδικασία, κατέφεραν να εξοικονομήσουν πολλά ε, χρήματα. Δεν πέρασε την πρώτη φορά η πρότασή μου για τον έλεγχο αυτό. Το υπέβαλα ξανά και υπήρχαν ε, αρκετές ε, οι ιστορίε που προέκυψαν. Παραδείγματο χάρη, το γεγονό ότι είμαστε στο Στρασβούργο μία εβδομάδα το μήνα και παρόλα αυτά υπάρχει φύλαξη από εταιρεία ασφάλεια όλο το χρόνο. Αν κοπεί αυτό και υπάρχει ασφάλεια μόνο στη διάρκεια της νοδολομελίας, ε, θα εξοικονομήσουμε ε, χρήματα. Τελικώς έγινε δεκτή η πρότασή μου για να γίνει ο έλεγχος ε, για τις εργασίες του Κοινοβουλίου, για τις υπηρεσίες ασφαλείας εγκρίθηκε η πρόταση και υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Το να εξοικονομήσουμε στις ταξιδιωτικές δαπάνες, ε, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πόσα χρήματα θα εξοικονομήσουμε. Εάν κάνουμε τον έλεγχο, θα μπορέσουμε να έχουμε και έναν έλεγχο της κατάστασης. Εγώ ελέγχω προσωπικώς ε, τα θέματα και τους τελευταίους 12 μήνα κατέφερα να εξοικονομήσω αρκετά χρήματα χωρίς ε, να κάνω κατάληξη των διοικητικών υπηρεσιών που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα έπρεπε λοιπόν να ακολουθήσουμε και εμείς την πρακτική των ελεγκτικών συνεδρίων, να κάνουμε τον εσωτερικό έλεγχο και να δούμε πόσα χρήματα θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσετε την ενδιαφέρουσα αυτή εμπειρία. Κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ θα ήθελα να εκφέρω τη γνώμη μου για δύο θέματα. Φυσικά εγώ ως φιλόλογος ε, βρίσκομαι σε αξιοζήλευτη θέση γιατί ομιλώ πολλές γλώσσες. Τώρα, και στην ε, συνεδρίαση ε, για τις σχέσεις με, την, με τους Τουρκοκύπριους συμφωνήσαμε να χρησιμοποιούμε δύο γλώσσες και νομίζω ότι έχεις μεγαλύτερες ε, επιτροπές χάρη οικονομίας θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την ε, διερμηνία και τη μετάφραση. Άλλωστε οι περισσότεροι από εμά ομιλούμε θαυμάσια αγγλικά. Άλλοι μιλούν ε, πολύ ωραία γαλλικά. Και στις καμπίνες διερμηνίας συνήθως η γλώσσα για το ρελέ είναι τα αγγλικά. Πολλές φορές εγώ μιλάω όταν μιλάω γερμανικά, όσοι δεν έχουν γερμανικά τα παίρνουν από τα αγγλικά. Και φυσικά τρέφω μεγάλο σεβασμό στο καθεστώ τη πολυγλωσία Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό καθένα να μπορεί να εκφράζεται και να διαβάζει στη μητρική του γλώσσα, αλλά χρειαζόμαστε κάποια ελαστικότητα στι πολιτικέ μα δεδομένων των τεράστιων οικονομικών δυσχεριών που αντιμετωπίζουμε. Να προσαρμόσουμε και τη δική μα νοοτροπία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά έξοδα για όλους μας ε, θα ήταν δυνατόν ε, να, να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις ώστε να βρούμε τα πιο οικονομικά ταξίδια. Θα μπορούσαμε και μόνοι μας να ψάχνουμε στο διαδίκτυο και να μην χρειάζεται υποχρεωτικά να προσφεύγουμε στο ταξιδιωτικό πρακτορείο που δεν δίνει και τις καλύτερες τιμές. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκαθάριση των εξόδων των αποστολών να δούμε πόσο κοστίζει το ταξίδι και ποια είναι η σχέση με την προηγούμενη εκαθάριση. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κατά αποκοπή ποσό και μετά τη διαφορά να την καλύπτει ο Ευρωβουλευτή, αν θέλει τα ταξίδια του να είναι πιο ακριβά ή ε, να επεκτείνονται και σε άλλα μέρη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ λογική πρόταση. Ο Γκέρον Φέρμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ντέρεκ Βόνο, ε, σκιώδης ηγητής, μίλησε εξ ονόματος της ομάδος. Ε, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάποια στοιχεία. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλησιάζουμε πλέον ε, σε συμφωνία για τα θέματα αυτά. Βέβαια, διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες και δεν έχουν επιληθεί όλα, αλλά είναι καλή η συνένεση στην οποία έχουμε καταλήξει. Ο κ. Φερνάνδε είπε ότι μπορεί να υπάρξουν κάποια νομικά προσκόμματα με τι τροπολογίε που προτείνουν το πάγωμα των δαπανών των ε, μελών και των διαφόρων επιδομάτων. Υπάρχει μία επιστολή από τον ε, πρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι η αρμόδια επιτροπή για το καθεστώ των ε, μελών, Συμφωνώ ω προ το μισθό. Κανένα δεν έχει το δικαίωμα να αγγίξει του μισθού μα. Αλλά για τη μείωση των δαπανών είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Επαφείτε βέβαια σε εσά, κύριε Πρόεδρε, να θεωρήσετε παραδεκτέ ή μη παραδεκτέ τι τροπολογίε αυτέ λόγω των προτάσεων τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Κατά μέσα ήταν ιδιαίτερα περίεργο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Προεδρείο έχει δικαίωμα να αποφασίζει ε, την ε, τιμολόγηση των επιδομάτων και θα αναλάβει καθήκοντα από ε, αυτούς που καθορίζουν τα επιδόματα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι νομικός δυνατό αυτό, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Αν για νομικούς λόγους δεν μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες για το πάγωμα των επιδομάτων, θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Θα πρέπει να το δούμε και να το επιλύσουμε. Για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας τώρα. Ζητήσαμε αρκετά πράγματα για να διευκρινιστεί η κατάσταση. Το βασικό ήταν ότι ζητήσαμε μια νομική βάση και έχει δίκιο η συγητής. Δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από τις αποφάσεις που ελήφθηκαν, ελήφθησαν πριν από το καλοκαίρι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν λάβαμε τις αποφάσεις αυτές για τις εκτιμήσεις, δεν γνωρίζαμε ποια ήταν η νομική βάση και ποιες ήταν οι συνέπειες της νομικής βάσης. Αυτά πλέον είναι γνωστά. Προτείναμε μια νομική βάση, αλλά θέλουμε και συγχρηματοδότηση από τα άλλα θεσμικά όργανα. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονό ότι η νομική βάση που προτείνει ο Γενικό Γραμματέα αποκλείει τη συγχρηματοδότηση από τα άλλα θεσμικά όργανα, γιατί τα άλλα ε, ε, θεσμικά όργανα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας, να χρηματοδοτήσουν συγγνώμη, το δικό μα κέντρο επιστογεπτών. Επομένω, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει συγχρηματοδότηση, όπω είναι και το να έχουμε την κατάλληλη νομική βάση. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε ποια νομική βάση μια επιτρέπει συγχρηματοδότηση από άλλα θεσμικά όργανα, να καταλήξουμε σε μια μια λύση από αυτού, αλλιώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα ω έχει. Ως προς τις ταξιδιωτικές δαπάνες, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό το Προεδρείο να κάνει μια πρόταση για τις λεπτομέρειες είναι αδύνατον για μας να ασχοληθούμε με θέματα όπως ε, το κατά πόσον ε, μας επιτρέπουν οι κανόνες να ταξιδεύουμε σε θέση business ή οικονομική, αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάρτες μιλίων, ε, συχνών ταξιδιωτών και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση για όλες αυτές τις λεπτομέρειες από πλευράς Προεδρίου και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Στον κύριο Ρικέ να πω το εξής. Έχουμε δύο τροπολογίες που προτείνουν κάποιες λύσεις για το θέμα αυτό. Καταρχάς μια συγκριτική μελέτη για τα εθνικά κοινοβούλια. Ναι, έχουμε καταθέσει τροπολογία για να κάνουμε συγκριτική μελέτη με τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να καταλήξουμε σε καλές ιδέες για περιττέρου εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και να έχουμε και μια εικόνα του κόστους ε, των άλλων κοινοβουλίων. Είναι υπερβολικές οι δικές μας οι δαπάνες σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόκειται λοιπόν για πρόταση η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Για το Γραφείο Ταξιδίων. Συμφωνούμε με τον κύριο Ρικέ και τον κύριο Άλβαρο ότι υπάρχουν προβλήματα με το Γραφείο Ταξιδίων. Επομένως, προτείνουμε το Προεδρείο να εξετάσει αναθεώρηση της συμφωνίας με το Γραφείο Ταξιδίων ε, και να δούμε τι προβλήματα προκύπτουν. Και τώρα πρέπει να μιλήσω με τον άλλο μου ρόλο. Δεν θα πρέπει να μιλώ εξ ονόματο τη πολιτική μου ομάδα, αλλά εξ ονόματο τη Σουηδική Αντιπροσωπεία η καλύτερη λύση θα ήταν να υπάρχει μία έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα δώσει απευθεία δυνατότητα για τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων. Πολλά μέλη κατέθεσαν τροπολογία προ αυτή την κατεύθυνση και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Τώρα όμω μιλώ μόνο εξ ονόματο του υποφαινόμενου και όχι εξ ονόματο τη ομάδα μου. Ευχαριστώ. Είχαμε προβλήματα μετάφραση. Την τελευταία σα πρόταση τη χάσαμε. Ο Γιάνν Μίλτερ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα διαπιστώσετε, σπάνια μιλώ τη γλώσσα μου. Συνήθως στις, επι... στις επιτροπές χρησιμοποιώ αγγλικά, γιατί πιστεύω ότι στα πολιτικά ο στόχος είναι να πείσουμε τους άλλους και πιστεύω ότι οι περισσότεροι ε, μιλούν αγγλικά, οπότε έχω μια μικρή ελπίδα ότι είμαι πιο πιστικό στα αγγλικά από ό,τι στα ολλανδικά. Βέβαια αυτό προς απογοήτευση των διερμηνέων. Πάντω όντω, σε πολλές συνεδριάσεις δεν χρειάζομαι διερμηνία. Τώρα κάτι άλλο. Πριν από εδώ και δύο-τρία χρόνια έχουμε το σύστημα του Webstream. Αν δεν κάνω λάθος και η σημερινή μας συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω του Webstream και άρα όλοι οι λαοί της Ευρώπης μπορούν να μας ακούσουν. Αν τώρα σε μια δημόσια συνεδρίαση ακυρώνουμε μια γλώσσα για την οποία επενδύσαμε και μέσω του Webstream, το Webstream γίνεται άχρηστο γιατί δεν αναμεταδίδεται στη συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό να το έχουμε υπόψη στις δημόσιες ε, συνεδριάσεις. Και με τις επενδύσεις που κάνουμε και με την ελπίδα ότι πολλοί συμπολίτες μας παρακολουθούν, δεν έχουμε βέβαια καμία ένδειξη γι' αυτό, καμία απόδειξη, αλλά ελπίζουμε ε, να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει αναμετάδοση μέσω του webstream σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ, Νέλα. Σε τέτοια περίπτωση θα ισχύει το ίδιο με αυτό που ισχύει για την επίσημη εφημερίδα και για την ανάγνωση του γραπτού κειμένου των πρακτικών δηλαδή των δημόσιων συζητήσεων. Το κείμενο αναγράφεται στη γλώσσα του ομιλητή, οπότε όποιος γνωρίζει αυτή τη γλώσσα μπορεί ε, να διαβάσει, ενώ οι άλλοι όχι. Ράινερ Μπέγκε. Σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ βουλευτών και όπου ζητείτε θα πρέπει να διατίθεται πλήρως και διερμηνία και μετάφραση. Βέβαια είναι και σημαντική πολυτέλεια αυτή που προσφέρουμε εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό ευχαριστώ οι συγητές και οι συγητές που κατόρθωσαν να θέσουν το θέμα αυτό και με εντατικό τρόπο μάλιστα στις συζητήσεις με το Προεδρείο κάτι που αποτελεί και απόδειξη ότι έχουμε και πολλές δυνατότητες να δείξουμε στην κοινή γνώμη ότι πηγαίνουμε σε ένα περιθώριο 1,9 και λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη για εξοικονομήσεις και μέσα στον ίδιο προπολογισμό. Μπορούμε να δούμε κάποια άλλη στιγμή πώς συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ανάγκη να μάθουμε όλοι αγγλικά γιατί ε, στους εθνικούς προϋπολογισμούς παιδείας ε, τους βαρύνει αρκετά η εκμάθηση της Αγγλικής. Το πακέτο στο σύνολό του βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ένα πράγμα θέλω να τονίσω ακόμη. Θυμούμε ότι χρειαστήκαμε πάνω από μια δεκαετία για να εξεύρουμε λύση σε διαθεσμικές ε, διαπραγματεύσεις αλλά και εδώ στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα, να κάνουμε ορισμένες μεταρρυθμίσεις και σε σχέση με το καθεστώ των βουλευτών και σε σχέση με τη χρηματοδότηση των συνεργατών και βεβαίω και για άλλα θέματα. Όποιο όμω τα ξαναρχίσει, τα ξανανοίξει όλα αυτά, ανοίγει την πηξίδα τη Πανδώρας και τίθεται και νομικά προβλήματα πρέπει να λυθούν σοβαρά υπόψη και που δεν μπορεί απλώ κανεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική σχέση μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπή Προπολογισμών, εγώ πιστεύω ότι οι επιτροπέ πρέπει να κάνουν τη δουλειά του στο παρελθόν όταν ήμουν εκεί στην θέση σου, αλλά συχνά εξοργίστηκα διότι το Προεδρείο δεν είχε πράξει το καθήκον του και εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμών αναγκαστήκαμε να αναλάβουμε τις ε, ευθύνες μας και στην Ολομέλεια και στη συνεδρίαση και κατορθώσαμε με εντατικό διάλογο με το Προεδρείο να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Εξακολουθώ και είμαι της ιδέας ότι πρέπει να τηρείται ο κανονισμός του σώματος. Αν όμως κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του μέσα στο κοινοβουλίο τότε προκαλείται ένα κενό. Και εκεί βέβαια πρέπει να παρέμβει εντονότερα η Επιτροπή Προϋπολογισμών όταν τη δουλειά του δεν κάνει το Προεδρείο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια εύλογη ισορροπία που πρέπει να εξευρεθεί. Εάν τεθεί το θέμα των μισθών, γιατί ο βουλευτής να αμείβεται με το 38,5% του μισθού του Ευρωπαϊκού Δικαστή, του Ευρωπαϊκού Δικαστή, συγγνώμη. Φαίνεται πως αξίζουμε μονάχα το 1 τρίτο. Επίσης, ορισμένοι βουλευτές καλούνται να πληρώσουν και εθνικούς φόρους, όχι σε όλες τις χώρες μέλη ωστόσο. Για μας τους Γερμανούς βουλευτές λοιπόν καλούμαστε να πληρώσουμε 700 1000 ευρώ παραπάνω φόρο. Όσο λοιπόν δεν ε, υπάρχει ισοτιμία εκεί, δεν θα δεχθώ και εγώ τροπολογίες άλλων συναδέλφων οι οποίοι δεν υφίστανται το ίδιο καθεστώς. Και όταν μιλούμε και για την, ε, τα, ποσό, τα ποσό κατά αποκοπήν, πρέπει και αυτό να συζητηθεί πάλι υπό το φως της ισότητας των βουλευτών. Ας μην λησμονούμε ότι υπάρχουν εδώ βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν 200.000 ε, ψηφοφόρους και άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούν ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους όπου χρειάζεται πολύ διαφορετική εργασία στην εκλογική περιφέρεια. Ας μην υπεραπλουστεύουμε λοιπόν τα πράγματα παίρνοντα την ε, μηχανή του κουρέματος του γκαζόν και κάνοντας τα όλα ίδια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έξοδα ταξιδιών. Τα γραφεία μας μπορούν να αναλάβουν τη δουλειά αυτή. Δεύτερο, business ή economy flex, εισιτήρια δηλαδή. Νομίζω ότι εδώ είναι περιττή η διαφωνία διότι υπάρχουν ορισμένε περιπτώσεις όπου πρέπει κανείς να ταξιδέψει στην business class. Εγώ βλέπω άλλο θέμα. Ωραία είναι τα ταξίδια των αντιπροσωπιών και σίγουρα έχουν μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά για εξετάστε λίγο το κόστος εκεί. Εκεί μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον να εγγύψουμε σε αυτό, στη μελέτη αυτού του κόστους και τώρα, σε μια περίοδο όπου αμφισβητείται ολόκληρη η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως οι συνάδελφοι θα έπρεπε να κινητοποιηθούν περισσότερο στις εκλογικές τους περιφέρειες και να ταξιδεύουν λίγο λιγότερο ανά τον κόσμο. Και μην λησμονούμε ότι η παράταση της εργάσιμης εβδομάδας θα έχει κάποιο κόστος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε βουλευτής θα είναι παρόν στην, ε, στις Βρυξέλλες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, μπορεί να είναι μόνο από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, διότι θα είναι εδώ αναλόγως με το πότε συνεδριάζει η Επιτροπή του. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους ώστε τα πράγματα να παραμείνουν μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μια λογική εξέλιξη εν το συνόλο. Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να συζητήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες ακόμη, όπου μπορούμε να καταδείξουμε νομίζω και σε, κάποιες, συμβασμού. κάποιους συμβασμούς. Ταυτόχρονα όμως μην δυσμονώντας και τα κελεύσματα της κοινή λογικής. Η ώρα προχωρεί. Έχουμε τον Σαλβατόρ Καρίγκα και δύο συναδέλφους που ήδη ζήτησαν το λόγο και Ζήτησα να δευτερολογήσουν. Παρακαλώ, Σαλβαντόρ, να είστε σύντομο για να προλάβουμε να ξανακούσουμε και τον εισηγητή μας με τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια συνεδρίαση είχαμε, μετά με την Οικονομική και Κοινωνική Ένωση χαίρομαι που μπορούμε να έχουμε και μια Δημοσιονομική Ένωση μετά την ενοποίηση της δημοσιονομικής αντιμετώπισης των Ευρωβουλευτών πρότεινε ο κ. Μπέγκε. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν πραγματικά σημαντική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση, μια τέτοια φορολογική ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που ήδη ανέκυψαν στη συζήτηση. Καταρχήν πιστεύω, δεν πιστεύω ότι εξορθολογισμός των δαπανών της διερμηνίας θα οδηγήσει σε μείωση της διερμηνίας. Απλώς θα κάνουμε μια καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και θα τους χρησιμοποιήσουμε εκεί που χρειάζονται. Εμείς οι συντονιστές έχουμε πολλές συνεδριάσεις εκτός των επίσημων αιθουσών και γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα χρήσιμη η διερμηνία, αλλά μερικέ φορέ εκεί που τη χρειαζόμαστε δεν έχουμε. Προτείνουμε λοιπόν μια καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, πιο αποτελεσματική και δυνατόν και πιο φθηνή. Σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά έξοδα, η πρόταση Φερνάντε είναι πολύ λογική, γιατί λαμβάνει υπόψη ένα τμήμα των προτάσεων που είχε καταθέσει το ΕΛΚ και λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις των σοσιαλιστών, των φιλελευθέρων και των πρασίνων. Νομίζω ότι είναι αρκετά συνενετική αυτή η πρόταση. Και πρώτα απ' όλα είναι συνενετική, συνενετική γιατί είναι ισορροπημένη. Γιατί άλλε προτάσεις, για παράδειγμα του κυρίου Πόρτας, είναι διακριτικέ. Είναι πολύ αυθαίρετη αυτή η διάκριση ε, ως προς τις ώρες του ταξιδιού και δεν αφορά ή δεν καλύπτει για παράδειγμα τα ταξίδια που γίνονται με αυτοκίνητο ή με τρένο. Γιατί να μην περιληφθούν και αυτά. Επίσης ε, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών καταστάσεων. Το μόνο που κάνει ο κύριος Πόρτες είναι να προτείνει διακριτική μεταχείριση. Νομίζω ότι η πρόταση του κύριου Φερνάντες είναι πιο λογική και ισορροπημένη. Σε ό,τι αφορά το πάγωμα των ημερήσεων αποζημιώσεων. Στην συνδιαλλαγή που είχαμε το πρωί κατάλαβα ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου. Το Προεδρείο δηλαδή καθορίζει το επίπεδο της να αναπροσαρμογής ε, ή της αύξησης των ημερήσεων αποζημιώσεων. Εμείς μπορεί να έχουμε πολιτική εντολή, να δώσουμε μια πολιτική εντολή ή να κάνουμε ένα αίτημα προς το Προεδρείο ζητώντας πάγωμα των ημερήσεων αποζημιώσεων, αλλά στη τελική ανάλυση το Προεδρείο είναι αρμόδιο να καθορίσει το ποσοστό αναπροσαρμογής αύξησης. Τώρα, αν δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο θέλει να παγώσει τι ημερήσει αποζημιώσει στο επίπεδο του 2011, τότε το Προεδρείο δεν θα εφαρμόσει αυτή την τήσια αύξηση, αλλά θα εκπληρώσει την πολιτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά κατάλαβα από την πρωινή συνδιαλλαγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον οίκο τη Ευρωπαϊκής Ιστορίας, πιστεύω ότι στη διάρκεια τη πρωινή συνδιαλλαγή που είχαμε, τα πράγματα ήταν ε, καθαρά και σαφέστατα. Υιοθετήθηκε μια νομική βάση και ήταν απαραίτητη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η συγχρηματοδότηση. Αυτό που είπαμε το πρωί στη συνδιαλλαγή, αυτό που μας είπε ο, Βε, ο Γενικός Γραμματέας το πρωί για τον Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, είναι να δούμε πώς θα ε, εμπλέξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια παροχή υπηρεσιών. Και είπε ότι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι την παροχή περισσότερων συνήθω την κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένη περίπτωση όμω του Ευρωπαϊκή Ιστορία θα μπορούσε κάλλιστα να εξεταστεί μια διαφορετική αντίθετη ε, πρόταση, όπου την παροχή υπηρεσιών θα την παρέχει, ε, θα την προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υλοποιώντα αυτή τη χρηματοδότηση, την οποία συμφωνούμε όλοι. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κύριε Πόρτας, παρακαλώ, μία πρόταση μόνο. Και με μικρόφωνα γίνεται. Λακανικά, μόνο μία παρατήρηση έχω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπέγκε. Μία και μόνο τροπολογία υπάρχει από όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί που αφορά άμεσα το καθεστώς του βουλευτού. Είναι δική μου αυτή η τροπολογία και προτείνει το πάγωμα των μισθών. Όντως, η τροπολογία αυτή εμπίπτει στο άρθρο 10 που προβλέπει ότι ο μισθός του βουλευτή είναι 38,5% του μισθού δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή και μόνο στην περίπτωση αυτή θα χρειαζόταν ένα πολιτικό μήνυμα δικό μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να γίνει διάλογος με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συμφωνία ή να τροποποιήσουμε το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 10 του καθεστώτος του βουλευτού ή να καταλήξουμε σε μια γενική συμφωνία που θα παγώνει το, το σύνολο των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρα 40, 50, 100 δικαστές. Αυτούς θα αφορά. Και νομίζω ότι πολύ πιο εύκολο είναι να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία από ότι αυτό που, επιδιώκει το Συμβούλιο. Να τροποποιήσει δηλαδή άρθρα της ίδιας της συνθήκης Λισαβόνας που κανονικά είχαν προβλεφθεί να ισχύουν για 30 χρόνια. Και αυτό, αυτό κάνει το Συμβούλιο ουσιαστικά. Καμία, κανένα κουτί της Πανδώρας δεν πρόκειται να ανοίξουμε είναι μια πολιτική πρωτοβουλία που αφορά ένα συγκεκριμένο άρθρο του καθεστώτος του βουλευτού. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης αν θα το επιχειρήσουμε ή όχι. Όλα τα υπόλοιπα σημεία, ταξιδιωτικά έξοδα, γενικά έξοδα, επιδόματα, ημερήσεις αποζημιώσεις, όλα αυτά είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου. Και αυτό που θα ήταν ε, από εμά αναμενόμενο είναι να εκφράσουμε την προθυμία μας να προβούμε σε περικοπές όχι μόνο στη λειτουργία, αλλά οφείλουμε να κάνουμε κάποιες περικοπές και στην ίδια τη διάρθρωση των δικών μας αμοιβών. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ, το καταλάβαμε κύριε Πόρτας. Ένα λεπτό και ο κύριος Ρικέ. Μία ερώτηση. Το θέμα το γλωσσικό είναι πολύ σημαντικό. Ε, υπόψη και η προσθήκη μιας νέας γλώσσας. Ε, συμπεριλήφθηκε και αυτό στην ανάλυση σας. Πολύ ωραία. Ναι. Ο Ράιμερ, μισό λεπτό να απαντήσει στον κύριο Πόρτας. Προσοχή, μην θίξουμε τα πολύ πτυχα θέματα του καθεστώτος των βουλευτών, διότι αποτελεί την πηξίδα της Πανδώρας. Μέσα σε όλο το δόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 16.000 πρόσωπα τα οποία κερδίζουν περισσότερα από τους ευρωβουλευτές. Αν ανοίξουμε λοιπόν τώρα και πάλι την υπόθεση του καθεστώτος του ευρωβουλευτού θα καταλήξουμε πάλι σε μια συζήτηση ανάμεσα στο ότι πρέπει εμείς να ε, βάλουμε τα, να καθορίζουμε μάλλον τους μισθούς ε, του Ευρωβουλευτού, όπως τις αμοιβές μάλλον, όπως ε, γίνεται και στις Εθνικές Βουλές και ανάμεσα στις επικίνδυνες άλλες απόψεις. Δεν προωθεί την υπόθεσή μας μια τέτοια συζήτηση και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου ένα πράγμα είναι σαφές και σημαντικό. Το βασικό μήνυμα θα πρέπει να είναι και του εισηγητού μας και του σκιώδου εισηγητού που καταφέραμε να διατηρήσουμε το 3,2% στο σύνολο του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο μήνυμά μας. Και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε καταφέρει πολλά. Και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσα στο σώμα, θα έχουμε δυνατότητες και τα επόμενα χρόνια που θα πρέπει με συνέπεια να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Φάρμε ένα λεπτό. Για το καθεστώς των βουλευτών. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Μπέγκε σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Να μην τις αγγίξουμε. Δεν μπορούμε να τις τροποποιήσουμε με τροπολογίες του προϋπολογισμού. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως την, ε, την αριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων, δεν συμφωνώ διότι βασισόμαστε στο 38,5% αλλά δεν ε, μας υποχρεώνει το καθεστώς των βουλευτών να κάνουμε τη μαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων. Εμείς καθορίζουμε τα ποσά στα κονδύλια του προϋπολογισμού και δεν νομίζω ότι είναι προνόμιο του Προεδρείου που μπορεί να αναλάβει δηλαδή να καθορίζει αυτό τα ποσά αυτά. Εγώ θα ήθελα εσείς κύριε Πρόεδρε να το ελέγξετε. Συμφωνώ ε, για τι αποζημιώσει, αλλά για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν είμαι βέβαιο. Νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε, διότι έχουμε έναν αριθμό ε, ε τροπολογιών που ζητούν πάγωμα των επιδομάτων. Εμεί ζητούμε πάγωμα όλων των επιδομάτων και των ημερήσιων αποζημιώσεων και των γενικών επιδομάτων και όλων. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε ω Επιτροπή προπολογισμών. Και ασφαλώς υπάρχει διαφορά ανάμεσα στι αποζημιώσει, δηλαδή στι αμοιβέ και στην τιματική αναπροσαρμογή. Τέλος η κυρία είναι και μετά πρόταση του εισηγητού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήρθα με κάποια καθυστέρηση, ήμουν στη διάσκεψη των ε, Προέδρων και επαναλαμβάνω τώρα αυτό που είπαμε και σήμερα το πρωί στην ε, Επιτροπή Συνδιαλλαγής που είχαμε με το Προεδρείο. Ζητήσαμε από το Προεδρείο κάποιες μελέτες για κάποιους τομείς ε, δαπανών, όπως για παράδειγμα την ανάγκη να υπάρχει περισσότερο προσωπικό λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας και πολλά άλλα, τα οποία ε, εξ όσων κατάλαβα δεν απαντήθηκαν ποτέ. Υπήρξαν κάποιες φήμες ότι το νέο καθεστώς σημαίνει και περισσότερες δαπάνες από πλευράς ταξιδίων και πάλι όμως δεν υπάρχει αξιολόγηση από αυτού και επομένως ε, εδώ και πάλι προκύπτει το ουσιώδες να γνωρίζουμε από πού προέρχονται, να έχουμε μελέτες για αυτά. Συμφωνώ με τα όσα ακούστηκαν για την νομιμότητα ή το παράνομο του παγώματος των ε, επιδομάτων Κατά την άποψή μου δεν τίθεται θέμα νομιμότητας. Υπάρχει μια επιστολή από την νομική υπηρεσία ε, η οποία μας υπευλήθη χθες και λέει ότι και ο μισθός και τα επιδόματα ε, έχουν νομικούς περιορισμούς ως προς το πάγωμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε με τη νέα νομική βάση, για την οποία παραπιπτόντως μόλις χθες άκουσα, να μπορούμε να έχουμε ε, διπηρεσιακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για λύση, διότι ούτως ή άλλως το κόστος θα βαραίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντί εμάς. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε εξοικονόμηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό στο σύνολό του. Η διπηρεσιακή συμφωνία λοιπόν κατ' εμέ δεν είναι λύση. Ευχαριστώ. Je vous remercie. Καλώ, ευχαριστώ. Πρόκειται για επιστολή τη ε, Νομική επιτροπή, όχι τη νομική υπηρεσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σχεδόν 12 η ώρα. Στι 12, σε 4 λεπτά, αλλάζει το καθεστώ διερμηνία στην συνεδρίασή μα. γιατί στι 12 αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών. Θα έχουμε κάποιε γλώσσε, αλλά όχι όλε τι γλώσσε. Οπότε στρέφομαι προς τον εισηγητή μας. Για το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2012, μετά τη συνδιαλλαγή και την παρουσίαση των συμπερασμάτων τη της συνδιαλλαγής, είχαμε κύριε εισηγητά μια πολύ πλούσια και γεμάτη ανταλλαγή απόψεων. Τι θέλετε, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τώρα ή να ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών για να το συζητήσουμε μεταξύ μας συντονιστές. Καλύτερα έτσι. Οπότε, οι, οι συντονιστές συνεδριάσουν 12 με 2 με λιγότερες γλώσσες οπότε θα διακόψω εδώ παρακαλώντας όσους δεν συμμετέχουν στους συντονιστές να εγκαταλείψουν την αίθουσα και θα επανέλθουμε στις 3 με την κανονική μας συνεδρίαση. Λύεται η συνεδρίαση η τακτική, να παραμείνουν παρακαλώ στην αίθουσα μόνο οι συντονιστές.